Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Θα ήθελα να καλωσορίσω απευθείας τον στονό Υπουργό Οικονομικών, τον Ντόμας Τόμιστε, ο οποίος δέχτηκε ευγενικά την πρόσκλησή μας να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της Εστονικής Προεδρίας στον τομέα των οικονομικών και νομισματικών θεμάτων, τα οποία νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Μία παρατήρηση παρακαλώ. Είναι απαράδεκτο να ξεκινάει η συνεδρίαση με 20 λεπτά ε, καθυστέρηση. Συστηματικά καθυστερούμε. Υπάρχει κόσμο που περιμένει εδώ, εδώ και 25 λεπτά να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Και ο ε, καλεσμένος μας. Παρακαλώ, θα ήθελα να ζητήσω από τον Πρόεδρο και τη Γραμματεία να μην επαναληφθεί. Ο πρόεδρο. έχετε δίκιο βεβαίω. Ε, εγώ είχα κάποιο πρόεδρα και πρόβλημα και καθυστέρησα ένα τέταρτο και ζητώ συγγνώμη αλλά μπορείτε να δείτε από τα πρακτικά μας ότι δεν συμβαίνει συστηματικά αυτό. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Έλεγα λοιπόν ότι η Εστονική Προεδρία συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχή διαπραγμάτευση πολλών ε, σημαντικών ε, νομοθετικών ε, θεμάτων στο προηγούμενο εξάμεινο. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον Πρέσβη και όλη την ομάδα η οποία με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα συνέβαλε στην πρόοδο των εργασιών μας στον τομέα αυτό και θα ήθελα να υπενθυμίσω τρία σημαντικά θέματα, τα οποία ε, απεδείχθηκαν ιδιαίτερα περίπλοκα και καταφέραμε παρόλα αυτά να έχουμε πολύ ικανοποιημένα αποτελέσματα και χρονικά αλλά και ως προς τα αποτελέσματα. Το πρώτο θέμα ήταν ιδιαίτερα περίπλοκο, είχαμε καθυστερήσει στο Συμβούλιο, αλλά τελικά καταφέραμε να σεβαστούμε τις προθεσμίες μας και κυρίως ε, να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Έχουμε και την ταχεία διαδικασία που πραγματικά αποτέλεσαν και δοκιμή. Είδαμε τι ακριβώς ε, γίνεται και τα καταφέραμε. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα και χαίρομαι που η Εστονική Προεδρία διαδραμάτισε κομβικό ρόλο διότι ε, είχαμε και ε, θετικά αποτελέσματα στην οδηγία για την ε, καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων ε, για το ξέπλυμα χρήματος. Ξέρετε ότι ήταν κάτι το οποίο καθυστερούσε μήνες και η κάθε προεδρία συνέβαλε μεν στις εργασίες, αλλά δεν καταφέρναμε να ολοκληρώσουμε. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση. Πολλοί αμφισβητούσαν ακόμα και το ενδεχόμενο να κλείσει το θέμα αυτό και παρόλα αυτά τα καταφέραμε και μάλιστα με πολύ καλό τρόπο και καταφέραμε να έχουμε στην Ευρώπη το προηγμένο ε, καθεστώς ε, καταπολέμησης νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων ε, στον κόσμο. Να συγχαρώ λοιπόν την Προεδρία, θα μας τα πει βεβαίως και ο Υπουργός. Δεν ασχολούμαστε μόνο με τους τριμερείς διαλόγους, αλλά γενικότερα με τα υπόλοιπα θέματα, τα οποία νομίζω ότι οδήγησαν και στην επιτυχία της Εστονικής Προεδρίας. Παρακαλώ, Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Ρομπέρτο. Θα μιλήσω αγγλικά. Ε, Συγγνώμη, θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα για να ακούσετε και την εστονική γλώσσα. Αξιότιμα μέλη, κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και πάλι. Σήμερα θα σας παρουσιάσω εν συντομία την πρόοδο που επιτύχαμε στα βασικά θέματα τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο των ε, θεματολογίων του ΕΚΟΦΗΝ ε, στη διάρκεια της Εστονικής Προεδρίας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια σύντομη επισκόπηση της οικονομικής κατάστασης. Το τελευταίο εξάμεινο η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συνέχισε να αυξάνεται ε, σταθερά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην πρόβλεψη του φθινοπόρου επιβεβαίωσε ότι το 2017 η οικονομική ανάπτυξη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ευρωζώνη θα υπερβούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτές οι θετικές τάσεις θα συνεχιστούν το 2018 και το 2019 παρά το γεγονός ότι θα πάνε με πιο βραδείς ρυθμούς. Επίσης, ε, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η ανάπτυξη βοήθησε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ε, το ποσοστό της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο χαμηλότερο ποσοστό του από το 2009. Η οικονομική ανάπτυξη συνέβαλε επίσης ε, στη μείωση των δημοσίων ελλημάτων. Το παρόν λοιπόν ε, ευνοϊκό οικονομικό πλαίσιο προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να συνεχίσουμε τις διαρθρωτικές βελτιώσεις των οικονομιών μας, καθώς επίσης και το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης. Και αυτό με οδηγεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ετήσια διαδικασία ε, συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη διάρκεια της Εσθονικής Προεδρίας, τον Οκτώβριο, το Συμβούλιο αξιολόγησε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2017. Ο στόχος της αξιολόγησης ήταν ε, να δούμε τι διδάγματα μπορούμε να αντιλήσουμε και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα ε, από τα κράτη-μέλη. Ε, η διαδικασία εξελίχθηκε συν το χρόνο στο εξάμεινο και έχει εξομαλυνθεί και είναι και πιο αποτελεσματική. Μία απόδειξη είναι το γεγονός ότι αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο βεβαίω είναι πιο σημαντικό είναι ότι τα αποτελέσματα της εφαρμογής των συστάσεων ε, είναι ακόμα κάτω των ε, προσδοκιών μας. Υπάρχει ακόμα αρκετό περιθώριο βελτίωσης και ιδιαίτερα ε, το γεγονός ότι πρέπει οι μεταρρυθμίσεις να αποτελέσουν κτήμα των κρατών μελών. Ελπίζω ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα εκτιμήσουν πόσο σημαντικές είναι οι συστάσεις που προτείνονται. Καταρχάς είναι προς το συμφέρον των κρατών μελών και ελπίζω ότι ότι ε, θα προσπαθήσουν όλοι να ε, κάνουν τις μεταρρυθμίσεις. Επίσης, ε, τα διδάγματα που αντλήσαμε ελπίζω να βοηθήσουν για περαιτέρω πρόοδο. Πρέπει να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και να βελτιώνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2018 ξεκίνησε ως συνήθως με την εξέταση της ετήσια έκθεση ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Συμβούλιο και επίση ε, την έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνηση και ε, το σχέδιο συστάσεων του Συμβουλίου για την οικονομική πολιτική τη Ευρωζώνη. Ολοκληρώθηκε η σύσταση για την Ευρωζώνη και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του ΕΚΟΦΗΝ εχθές στις 23 Ιανουαρίου και πλέον ε, μπορεί να την εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο. Οι φετινές ε, συστάσεις ε, ζητούν μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που υποστηρίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη και επικεντρωνόμαστε σε ισορροπημένα και δημόσια οικονομικά υψηλής ποιότητας με στόχο να αυξήσουμε την οικονομική ανθεκτικότητα. Επίσης, ζητάμε από τις χώρες Ευρωζώνης ε, να προσπαθήσουν να έχουν ε, μια ευρύτερα ουδέτερη ε, φορολογική στάση θέλουμε κατάλληλη διαφοροποίηση των δημοσιονομικών προσπαθειών ε, σε, στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, λαμβάνοντας υπόψη και το δημοσιονομικό χώρο και την ε, ε λύση προς τις άλλες χώρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ε, διασφάλισης της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών και της υποστήριξης της οικονομίας. Επιπλέον, οι ευνοϊκέ οικονομικές συνθήκε πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουμε κατάλληλα προστατευτικά μέσα ε, σε δημοσιονομικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύουμε και τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, από τις συστάσεις ε, γίνεται έκκληση προς τα κράτη-μέλη να υπάρξει πρόοδο ε, για την ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ένωση και τη οικονομική και νομισματική Ένωση οι πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και θα πρέπει να υπάρχει και εγγυημένη διαφάνεια για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Η πρόθεση των επενδύσεων είναι και βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από μια μακρά περίοδο στασιμότητας σε επενδύσεις, ε, πλέον οι επενδύσεις έχουν ξεκινήσει να ανακάμπτουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, κυρίως ε, λόγω ευνοϊκών οικονομικών συνθήκων και θετικών οικονομικών προβλέψεων, παρά το γεγονό ότι εξακολουθούν να είναι χαμηλές οι επενδύσεις του ιδιωτικού κλάδου. Ε, είμαι ικανοποιημένο που καταφέραμε να ξεπεράσουμε τι διαφορέ μα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόταση παράταση τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων μέχρι το 2020. Είναι μια ε, σωστή πρωτοβουλία. Αποδείχθηκε η προστιθέμενη αξία του ταμείου αυτού στη διάρκεια των πρώτων τριών ετών λειτουργίες και πιστεύω ότι θα αυξήσουμε τους στόχους επενδύσεων και θα έχουμε και επενδύσεις από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και έτσι το Ταμείο θα μπορέσει να γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο για να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις που χρειάζονται. Η συζήτηση για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ε, συνεχίζεται εδώ και αρκετό καιρό και έχουν προταθεί διάφορα πράγματα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Για να προχωρήσουν οι συζητήσεις για αυτό το κρίσιμο ζήτημα, η Εστονική Προεδρία οργάνωσε μία άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών στο Ταλίν τον Σεπτέμβριο και σε αυτή την άτυπη ανταλλαγή απόψεων ε, τέθηκαν τα θεμέλια για περαιτέρω συζητήσεις ε, στην ε, Σύνοδο του Δεκεμβρίου οι ε, εργασίες θα συνεχιστούν στις κατάλληλες συνθέσεις, και στο Eurogroup και στο ECOFIN. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο θα χρειαστεί υπομονή και χρόνο και θα πρέπει όμως να στοχεύσουμε σε κάποια απτά αποτελέσματα ε, βραχυπρόθεσμα. Έχει ήδη επιτευχθεί πρόοδο ε, σε μία σειρά από θέματα που αφορά την πρόοδο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ε, οι δέσμοι μέτρων για την Τραπεζική Ένωση και τις προτάσεις για την ε, Ένωση των Κεφαλαίων Η Τραπεζική Ένωση ήταν βασική προτεραιότητα της Εσθονική Προεδρίας. Πρόκειται για ένα ακόμα μακροπρόθεσμα πρόγραμμα, το οποίο απαιτεί και κοινό έδαφος ε, για πολλά αλληλένδετα, τεχνικά σύνθετα και ε, πολύ σημαντικά από πολιτική σκοπιά θέματα. Παρ' όλα αυτά υπήρξε καλή πρόοδος ε, για τη δέσμη μέτρων για τα τραπεζικά ζητήματα και περιλαμβάνονται μέτρα τα οποία θέλουν να μειώσουν τον κίνδυνο στο τραπεζικό τομέα. Όπως ε, συμφωνήθηκε στον οδικό χάρτη του Ιουνίου του 2016, Πρέπει να υπάρξει επαρκή πρόοδο για αυτές τις προτάσεις πριν ξεκινήσει η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ασφάλισης Καταθέσεων, που είναι βασικός πυλώνας της προτινόμενης αρχιτεκτονικής δομής της Τραπεζικής Ένωσης. Θα ήθελα να αναφέρω και δύο ε, νομοθετικές πράξεις οι οποίες ε, προχώρησαν με την ε, επίγουσα διαδικασία για να μειώσουμε τον κίνδυνο στον τραπεζικό τομέα. Καταρχάς μια οδηγία για την βαθμολόγηση των μέσων χρέους στις διαδικασίες αφαιρεγγιότητας, το, τη λεγόμενη ιεραρχία των τραπεζικών πιστωτών και επίσης ένα κανονισμό για τις μεταβατικές διατάξεις ε, για το IFRS 9 το διεθνές ε, λογιστικό ε, πρότυπο. Και τα δύο αυτά εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το Δεκέμβριο μετά από συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Οκτωβρίου οι ομάδες εργασίας του Συμβουλίου εξακολουθούν να επεξεργάζονται άλλες νομοθετικές προτάσεις που αφορούν την Τραπεζική Ένωση. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσει, ε, την οδηγία και τον κανονισμό, ε, την οδηγία για την ανακτήση ποσών και την επίλυση διαφορών σε τραπεζικό επίπεδο και τον κανονισμό για τον ενιαίο μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Ε, θα συνεχίσουμε τις τεχνικές συζητήσεις για αυτά τα περίπλοκα ζητήματα. Η, η οικονομική κρίση και η ύφεση η οποία προέκυψε στη συνέχεια ε, έχουν οδηγήσει σε τράπεζες, σε κράτη-μέλη με πολύ ψηλά επίπεδα ε, κόκκινων δανείων. Υπάρχουν κίνδυνοι για πιθανές ε, δηλήσεις και σε άλλες χώρες και μπορεί να αντιμετωπίσει και πρόβλημα ο τραπεζικός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε, ε, στην οικονομία στη, εν γέννη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Ιούλιο εγκρίθηκε ένα πρόγραμμα δράσης ε, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ε, δανείων αυτών στον τραπεζικό τομέα. Υπάρχει ένα μείγμα δράσεων πολιτικής για να μειώσουμε τον αριθμό των δανείων αυτών και να μην υπάρξουν αντίστοιχα φαινόμενα και στο μέλλον. Το Συμβούλιο επίσης συμφώνησε να αναθεωρεί το σύστημα αυτό τακτικά για να αξιολογεί πώς εξελίσσονται τα δάνεια αυτά στην Ευρώπη και ε, να δούνε και τι δράσεις έχουν αναλυφθεί και αν έχουν οδηγήσει σε αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή ε, προετοιμάζει μία δέσμη μέτρων για να εφαρμόσει το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής του Συμβουλίου για τα ε, δάνεια αυτά και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να βοηθήσει να επιτύχουμε τον κοινό μας στέχο, να μειώσουμε τον ε, ε, δημοσιονομικό κατακαιρματισμό και να διευκολύνουμε την ε, ροή κεφαλαίων εντός της ενιαίας αγοράς. Επιπλέον τα μέτρα αυτά μπορεί να έχουν και θετικά αποτελέσματα στη συζήτηση για τον επιμερισμό κινδύνου στον τραπεζικό τομέα, ιδίως όσον αφορά την προστασία για το SRF και το προτινόμενο πρόγραμμα ε, εγγύησης ε, ε, καταθέσεων, το οποίο συζητάται ακόμα στις τεχνικές εργασίες στο Συμβούλιο. Επιπλέον, Πέραν των όσων έκανε η Εστονική Προεδρία για την Τραπεζική Ένωση, υπήρξε και πρόεδρος για τα ε, όσα θα συνθέσουν την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Ε, προσπαθούμε να ε, μειώσουμε την εξάρτηση από τράπεζες και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για διαφοροποιημένες διόδους χρηματοδότησης. Οι ομάδες εργασίας του Συμβουλίου έκαναν πρόοδο όσον αφορά τα διάφορα θέματα που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Καταρχάς θα ήθελα να αναφέρω τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό της Υποδομής των Αγορών ο κανονισμός αυτός ε, θέλει να αυξήσει την ε, αναλογικότητα και να μειώσει το κόστος ε, για όσους συμμετέχουν, ιδιαίτερα για τους μικρότερους μετόχους και με την εκαθάριση των παραγόγων. Καταλήξαμε σε συμφωνία για την εντολή διαπραγμάτευση Συμβουλίου του Δεκέμβριου και το Συμβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει τον τριμερή διάλογο όταν θα είναι έτοιμο και το Κοινοβούλιο. Επίσης ξεκινήσαμε συζητήσεις για τις προτάσεις για την εποπτεία των ε, ε, κεντρικών αντισυμβαλόμενων σε τρίτες χώρες, καθώς επίσης και μία πρόταση για, ένα, ε, για πανευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά προϊόντα. Ε, αυτές οι συζητήσεις πιστεύω ότι θα επιτρέψουν στην Βουλγαρική Προεδρία να προωθήσει τις εργασίες αυτές περαιτέρω. Ένα άλλο σημαντικό θέμα στον τομέα αυτό αφορά τους ενισχυμένους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Καταλήξαμε στη συμφωνία για την οδηγία αυτή ε, σε περιβάλλον εμπιστοσύνης και καλή συνεργασία μαζί σα και με του συναδέλφου σα από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Η συμφωνία επετεύχθη τέλος Δεκεμβρίου και τώρα πλέον πρέπει να εγκρίνουν τη σχετική πράξη και τα δύο θεσμικά όργανα. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα στις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να προλάβουν τη χρήση ε, του ε, χρηματοπιστωτικού συστήματος για χρηματοδότηση ε, παράνομων δραστηριοτήτων. Η οδηγία επίσης θέλει να ενισχύσει τους κανόνες διαφάνειας για να μην υπάρχουν μεγάλης κλίμακας απόκρυψη κεφαλαίων. Και είναι τμήμα του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που εγκρίθηκε το 2016 μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη. Να ολοκληρώσω τώρα λέγοντας ε, δύο πράγματα για την φορολογία. Ένα από τα βασικά μας επιτεύγματα το τελευταίο εξάμεινο ήταν ε, η δημιουργία του ε, καταλόγου για τις ε, φορολογικές επικράτες οι οποίες δεν συνεργάζονται σε θέματα φορολογίας. Ο στόχος ε, ε, δεν είναι να είναι ο κατάλογος μόνιμος, στόχος είναι να αναθεωρείται τα επόμενα χρόνια και είμαι βέβαιος ότι η Βουλγαρική Προεδρία θα συνεχίσει με επιτυχία αυτές τις εργασίες βάσει της διαδικασίας που έχει καθοριστεί. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω την πρόκληση της ε, φορολογίας των εσόδων από την ψηφιακή οικονομία. Είμαστε βαθύτατα πεπισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση προκειμένου οι φορολογικοί κανόνες ε, να είναι κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή. Το Συμβουλίο Κοφίν του Δεκεμβρίου ενέκρινε συμπεράσματα για την φορολόγηση των εσόδων στην ψηφιακή οικονομία και είμαστε περήφαμοι που καταλήξαμε σε συμφωνία ε, για το ε, πακέτο ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ελπίζουμε ότι θα δώσει νέε πιθανότητε στου καταναλωτές και θα διευκολύνει το διασυνοριακό εμπόριο για τι μικρέ επιχειρήσει. Με αυτό ολοκλήρωσα την παρουσίασή μου. σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και προσβλέπω σε ερωτήσει σα.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 και για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με, την, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Θα δώσω τώρα στον κύριο Μπάλτς το λόγο να ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα και εγώ σε προσωπικό επίπεδο να σας ε, ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο η χώρα σας ε, Κάνει μια ε, προεδρία η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν εξαιρετική. Πρέπει να σας πω πως ήταν η πρώτη φορά που ασκήσατε την προεδρία του Συμβουλίου και η αλήθεια είναι πως οι τελευταίοι μήνες πραγματικά ήταν εντυπωσιακοί. Ένα σημείο είναι αυτό στο οποίο θα ήθελα εδώ να σταθώ και είναι μια σύντομη ερώτηση που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Μιλήσατε για την ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη. Ε, το ΕΚΟΦΗΝ να σας πω ότι χτες ενέκρινε τα συμπερίσματά του για την, χτες, για την ανάπτυξη, την ετήσια αυτή έκθεση και είπε πως η εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα έγινε σε επίπεδο προσπάθειας και δέσμευσης με μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα διάφορα κρατημέλη. Δηλαδή αυτό που μας είπατε εσείς είναι ότι μεν περνάμε μια πολύ θετική συγκυρία αυτή τη στιγμή, αλλά χρειάζεται και προσπάθεια για να πετύχουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Εντάξει, αλλά η δική σας χώρα ε, κάθε χρόνο ε, έχει εξαιρετικές επιδόσεις στις συστάσεις που γίνονται κράτος. Έχετε ένα έλλειμμα κάτω από το ε, οπότε η ερώτηση δική μου είναι η εξής. Πού βρίσκονται τα κλειδιά της επιτυχίας της χώρας σας και της κυβέρνησής σας. Πού αποδίδουμε αυτές τις εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Ξέρετε πως η τρέχουσα οικονομική συγκυρία επιτρέπει στις χώρες οι οποίες είχαν ενδεχομένως δυσκολίες ε, στο να ε, ισορροπήσουν τους προπολογισμούς τους, να ε, συγκεντρώσουν χρήματα στο αποθεματικό τους, να το πετύχουν και πρέπει να σας πω που η αστωνική προσέγγιση ε, ιστορικά μιλώντας ήταν πάντα η ίδια. Να υιοθετούμε κανόνες και όταν τους υιοθετούμε να συμμορφωνόμαστε όλοι με αυτούς. Γιατί μόνο τότε επιτρέπεται να συνεχίσουμε με την εισαγωγή νέων κανόνων. Αυτή είναι μια γενικότερη αρχή την οποία εμείς υπηρετούμε και θα ήθελα να σας εξηγήσω ε, τι συμβαίνει με την Εστονία και ποια είναι η εστονική προσέγγιση. Εμείς αυτό που έχουμε κάνει είναι να πιστεύουμε ότι τα δάνεια δεν ανήκουν σε αυτά που το έχει δανειστεί, αλλά σε αυτό που δανείζει. Και τα κόμματα, κυρίως στη δεξιά, έχουν προσπαθήσει ε, με ιδιαίτερη δυσκολία να φέρουν ισολογισμένους, ισοσκελισμένους ε, προϋπολογισμούς ε, και κατά τη διάρκεια της χρήσης χρησιμοποιήσαμε και τα αποθέματα που είχαμε στο αποθεματικό μας. Κάναμε τεράστιες περικοπές στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας και και μεγάλη χαρά διαπιστώνω πως η κοινωνία έδειξε κατανόηση. Έδειξε κατανόηση για την αναγκαιότητα αυτών των περικοπών. Και ακριβώς για το λόγο αυτό το εθνικό μας ε, αυτή τη στιγμή ο εξωτερικός δανεισμός ε, είναι κάτω από το 10% του ΑΕΠ και νομίζω ότι Είμαστε ε, στα χαμηλότερα επίπεδα στα 27 κράτη-μέλη και στον ε, ΟΣΑ και είναι πολύ καλά και τα αποθεματικά μας. Τώρα, μία από τις προτεραιότητες που δώσαμε είναι ε, να επανακινήσουμε την οικονομία μας. Και πρέπει να σας πω πως στην κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιήσαμε τα διαρθρωτικά ταμεία τα οποία χρησιμοποιήσαμε με το βέλτιστο δυνατόν τρόπο έτσι ώστε να μας βοηθήσουν να εισαγάγουμε τις τεράστιες αλλαγές που χρειαζόμασταν έτσι ώστε να αυξήσουμε τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Και βέβαια στηρίξαμε και την έρευνα και την τεχνολογία. Euh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Η χώρα σας έχει μία φήμη η οποία επαληθεύεται ότι έχετε στοιχηματίσει υπέρ της ψηφιακής οικονομίας και κάνατε και μία πολύ σημαντική διάσκεψη κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Και μάλιστα, όπως είπατε και εσείς, στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου εγκρίνατε και τα συμπεράσματα για τη φορολόγηση του ψηφιακού κόσμου. Όμως θα ήθελα να μου πείτε, με την εμπειρία που έχετε, συμφωνείτε με την εξή ιδέα, πως το ψηφιακό είναι κάτι το οποίο θα μεταλλάξει ε, όλη μας την οικονομία και είναι πολύ δύσκολο αυτή την ε, μετάλλαξη, την οικονομική, να τη συνδυάσουμε με μια φορολόγηση ε, του ψηφιακού κόσμου. Γιατί εμείς από την αρχή της ε, θητείας μας είπαμε η φορολόγηση θα πρέπει να είναι υπέρ της κοινωνίας αλλά με τρόπο που θα επιτρέπει την ανάπτυξη αυτή. Να επιστρέφει στην κοινωνία, με συγχωρείτε, με τρόπο που επιτρέπει την ανάπτυξη της οικονομίας. Τώρα, θα έχουμε ειδική ψηφιακή φορολόγηση για τις πλατφόρμες. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες εκεί και θα αφήσουμε στην άκρη τις προσπάθειες που θα έπρεπε να γίνουν εκεί που γίνεται η μάχη, που είναι ο εταιρικό φόρος, έτσι ώστε να ε, πληρώσουμε τα κενά και να προχωρήσουμε στην εγκαθίδρυση μιας πραγματικής ψηφιακή οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι όπως το λέτε. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, το θέμα της φορολόγησης των ψηφιακών ε, υπηρεσιών της οικονομίας ήταν ένα από τα θέματα τα οποία πιο πολύ συζητήσαμε και το οποίο είχαμε θέσει εμείς ως προτεραιότητα. Γι' αυτό και του δώσαμε τόση σημασία. Νομίζω πως η κοινή προσέγγιση της Ευρώπης, η κοινή κατανόηση του θέματος αυτούς στην Ευρώπη είναι πως Έχουμε κάποιες υφιστάμενες αρχές ε, για τα θέματα φορολογίας που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες και πως έφτασε η ώρα όλα αυτά να αναθεωρηθούν. Γιατί μέχρι σήμερα φορολογούσαμε βάσει της φυσικής παρουσίας, της φυσικής εγκατάστασης. Αλλά δεδομένων των ψηφιακών, της ψηφιακής τεχνολογικής πρόοδου, Μία εταιρεία δεν χρειάζεται να βρίσκεται σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, σε συγκεκριμένη χώρα. Μπορεί να βρίσκεται μέσα σε ένα iPad, σε έναν υπολογιστή. Οπότε, αυτό πολλές τίμιες εταιρείε που πληρώνουν τους φόρους τους τις βάζει σε μειονεκτική θέση. Γιατί φορολογούνται και οι ανταγωνιστές τους όχι. Με δράσεις και υπηρεσίες που προσφέρουν στην ίδια χώρα και παρόλα αυτά δεν φορολογούνται. Γι' αυτό καλωσορίζω ιδιαίτερα την γαλλική πρόταση για να βρούμε μια πιο γρήγορη λύση. Γιατί αν δεν καταφέρουμε σε επίπεδο όσα να βρούμε κάποια αποτελέσματα, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η βασική αρχή στο ΕΚΟΦΗΝ ήταν ότι θέλουμε μια παγκόσμια λύση που να βασίζεται ε, στην φορολογία έτσι όπως πληρώνεται σήμερα. δηλαδή στη φορολόγηση των εσόδων. Αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε βέβαια, θα πρέπει όλη μαζί η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τα κρατημέλη να προχωρήσει μόνοι. Αυτή η πλατφόρμα λοιπόν θα εισαχθεί ε, την άνοιξη στην σχετική συνάντηση που θα γίνει στον ΩΣΑ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λέρνερ. Η κυρία Λένερ, με συγχωρείτε, σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Η Εστόνια αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος της ψηφιοποίησης και καταλαβαίνετε ότι αυτό σας δίνει μια ευκαιρία στο να διαμορφώσετε τις προτεραιότητες στον ψηφιακό κόσμο. Είσαστε μία από τις πιο δικτυωμένες χώρες και είστε παράδειγμα για τους υπόλοιπους και για τα δημοσιονομικά σας, τι να πω, χρησιμοποιήσατε την ψηφιοποίηση και στρέψατε τους πολίτες στις δημόσιες υπηρεσίες μέσω ίντερνετ. Και νομίζω ότι αυτή ήταν μια εξαιρετική δυνατότητα που τους δόθηκε, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, έτσι ώστε να είναι οικονομικές ε, οι υπηρεσίε που προσφέρει το δημόσιο ακόμα και σε περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού. Όμως, σε ένα ψηφιακό κόσμο τι γίνεται όταν οι ψηφιακές υπηρεσίε χρειάζονται ειδικέ δεξιότητες και αυτές δεν υπάρχουν. Για παράδειγμα, ε, ξέρουμε τη γλώσσα, έχουμε smartphone, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε tablet. Μπορούμε λοιπόν αυτές τις υπηρεσίε να τις βρούμε στο διαδίκτυο. Εσείς τι κάνατε με αυτούς που δεν μπορούσατε, τους ηλικιωμένους για παράδειγμα, αυτούς που δεν έχουν τέτοιου είδους δεξιότητες. Αυτοί πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Εστονία επέλεξε να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές λύσεις, τα e-solutions, στο μέτρο του δυνατού. Και πρέπει να σας πω πως κερδίθηκαν χιλιάδες εργατόρες. Ε, βοηθήσαμε το φυσικό περιβάλλον, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί με τον τρόπο αυτό έχουμε διοικητικές διαδικασίες που είναι απλούστατες για όλους. Και θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Υποβολή φορολογικής δήλωσης. Ένα-δύο λεπτά παίρνει αν δεν έχεις πολλές επιπλέον πληροφορίες. Γιατί οι δικές μας φορολογικές υπηρεσίες έχουν ήδη προσυμπληρώσει το έγγραφο που κατεβάζεται διαδικτυακά, απλώς τσεκάρετε ότι είναι σωστό και το υποβάλλετε. Στόχος μας είναι λοιπόν οι επαφές με το κράτος ε, να είναι όσο το πιο εύκολες για τους πολίτες. Και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια πολύ ικανοποιητικά. Πράγμα που μας επιτρέπει όλους να συμμετέχουμε, αν θέλετε, στο ίδιο επίπεδο ε, πληροφοριών. Αυτό μας επιτρέπει, για παράδειγμα, να ε, υιοθετούμε ευκολότερα νομικές πράξεις και να τι κυρώνουμε φυσικά αργότερα. Υπάρχουν από εκεί και μετά μια σειρά από προγράμματα τα οποία εγγυώνται την προσβασιμότητα του διαδικτύου για όλους. Κατά τα τελευταία χρόνια, μία από τις προτεραιότητες μας αποτέλεσε η ευρυζωνική διαδικτυακή σύνδεση. Με άλλα λόγια, κάθε πρόσωπο, κάθε άτομο θεωρούμε η αποτελεί προτεραιότητα θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο. Είτε είναι νέος, είτε είναι ε, της τρίτης ηλικίας. Επίσης έχουμε μια σειρά από προγράμματα εκπαιδευτικά για εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν αποτελεί πρόβλημα για τους νέους γνωρίζουν φυσικά πώς να χειριστούν έναν υπολογιστή, αλλά είτε μας αρέσει είτε όχι, πέρα από τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες κρατικές ε, υπηρεσίες ε, θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει δυνατότητα για ηλικιωμένου ανθρώπους να μεταβαίνουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να λάβουν εκεί βοήθεια Πρόσφατο πρόσωπο. Ε. Κύριε σας ευχαριστώ. Και εγώ συμμερίζομαι την άποψη του Μπορχαμπάλς ότι η δική σας ε, προεδρία πράγματι στέφθηκε με επιτυχία για την Ένωση και θεωρώ πως το ζήτημα της ηγεσία, δηλαδή το πώς μπορεί να λάβει, να, να λάβει ένα ηγετικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει να κάνει με το μέγεθος της χώρας αλλά έχει να κάνει με τις ευέλτιστες ε, πρακτικές ε, και είδαμε για παράδειγμα η Φιλανδία έχει ηγετικό ρόλο στον εκπαιδευτικό τομέα, πως η Δανία έχει πολύ καλές επιδόσεις στην αγορά εργασίας, ε, πως οι κάτω το καλύτερο λιμενικό σύστημα και πως η Σουηδία ε, κατάφερε να βγει από την οικονομική κρίση μέσα σε ένα χρόνο χάρη σε μια ευρεία συνένεση εκεί. Οπότε σε ό,τι αφορά αυτή την επιτυχία έκβαση του προγράμματος ηλεκτρονικής εστονίας της ή εστονίας ε, ε, αυτό μας το παρουσιάζεται ως ε, αν θέλετε το πιο σημαντικό, την πιο σημαντική διάσταση από τη δική σας πλευρά οπότε θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω και ένα ακόμα ερώτημα ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη εναρμόνιση της φορολογικής βάσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί γνωρίζετε πως αποτελεί αυτό ακόμα ένα εργαλείο σε ό,τι αφορά την διαφοροποίηση ε, της οικονομικής οργάνωσης των διαφόρων κρατών μελών. Ε, όπως γνωρίζετε, ειδικότερα είναι σημαντική, αυτή, σημαντικό αυτό το εργαλείο για τις μικρότερες χώρες ε, προκειμένου να μπορέσουν να αναλάβουν και ηγετικό ρόλο σε διαφορετικούς τομείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματά σας. Ναι. Θεωρώ πως ε, πράγματι ε, κάθε κράτος μέλος της Ένωσης ε, έχει έναν τομέα στον οποίο έχει καταφέρει πολλά και βέβαια κάθε κράτος μέλος έχει τα δικά του προβλήματα. στην διάσκεψη του ΕΚΟΦΕΝ κάναμε μια σειρά από συζητήσει, ε, στο πλαίσιο των οποίων ε, τα διάφορα κράτη-μέλη αναφέρθηκαν στην πρόοδο που πέδιχαν σε ό,τι αφορά τον ε, τομέα τη παιδεία ή τον τομέα τη φορολογική μεταρρύθμιση. Και εκεί ακούσαμε δηλαδή την παρουσίαση των όσων πέτυχαν τα διάφορα κράτη-μέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κοινή φορολογική βάση για τις εταιρείε. Νομίζω πως ε, αφορά ο ζήτημα περισσότερο κάποιες ε, χώρες, κάποια κράτη-μέλη σε σύγκριση με άλλα. Ορισμένα δηλαδή κράτη-μέλη διστάζουν, φοβούνται να αλλάξουν το φορολογικό του σύστημα γιατί το θεωρούν ακριβώς ως επιτυχημένο ως ένα σύστημα που λειτουργεί καλά. Ενώ άλλα κράτη-μέλη θεωρούν πως θα πρέπει να προωθήσουμε ταχύτατα αυτήν την κοινή φορολογική βάση. Η πρόοδος που έχουμε επιτύχει στο δομέα των ε, ηλεκτρονικών υπηρεσιών ε, είναι εξαιρετικά σημαντική για μας και έχουμε αναπτύξει και το σύστημα EU Residency διαμονής δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο βοήθησε ε, στη μείωση της γραφειοκρατίας για τους ε, υπηκόους τρίτων χωρών έτσι ώστε να μπορούν και εκείνοι να συμμετέχουν στην ε, στονική οικονομία. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα σύστημα φοροαποφυγής, αλλά για ένα σύστημα δημιουργίας ή εδραίωσης κοινών κανόνων για όλους. Ευχαριστώ. Ο κ. Παπαδημούλης έχει το λόγο. Θα ήθελα και εγώ, κύριε Τόνιστε, να ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και να σημειώσω ότι και κατά τη γνώμη μου ο απολογισμός της Εστονικής Προεδρίας είναι θετικός. Θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο αφορά την ολοκλήρωση τραπεζικής ενοποίησης με την εγκαθίδρυση και του τρίτου πυλώνα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων. Είχατε στόχο να προωθηθούν μέτρα μείωσης του ρίσκου στον τραπεζικό τομέα. Και έχετε σε αυτό το θέμα ως απολογισμό κάποια θετικά βήματα. Η μείωση του ρίσκου μπήκε σε ένα δρόμο. Αλλά η αμοιβεοποίηση του ρίσκου παράλληλα που είναι απαραίτητη σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν για την ολοκλήρωση του τρίτου πυλώνα για να αποκτήσουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα εκατοστό του μέτρου. Και χωρίς τρίτο πυλώνα δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλοι οι οικονομολόγοι και η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λένε ότι τώρα πρέπει να προχωρήσει η ολοκλήρωση Τραπεζικής Ένωσης έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη να είναι πιο προετοιμασμένοι και πιο θωρακισμένοι αν αύριο υπάρξει μια κρίση, αν αύριο υπάρξει μια ύφεση. Τώρα που τα πράγματα είναι πιο ήρεμα, πρέπει να γίνουν τα βήματα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, πού βρέθηκαν οι δυσκολίες και τα εμπόδια και δεν προχωρήσατε καθόλου στο Συμβούλιο στον τομέα της παράλληλης αμοιβεοποίησης του ρίσκου. Ποια κράτη-μέλη είναι αυτά που βάζουν φρένο σε αυτό που έχει προτείνει η Κομισιόν, σε αυτό που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε αυτό που υποστηρίζει και ένα μεγάλο μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα θέλαμε μια ενημέρωση σε αυτό. Το δεύτερο θέμα αφορά στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Στη διάρκεια της Προεδρίας σας υπήρξε η μεγάλη αποκάλυψη των Paradise Papers, αυτό το σκάνδαλο της μέγα φοροδιαφυγής και είχαν προηγηθεί πριν από ένα χρόνο και τα Panama Papers. Επομένως η πραγματικότητα βοά ότι πρέπει να γίνουν βήματα εναρμόνισης, στενότερης συνεργασίας, αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης αυτής της μέγα φοροδιαφυγής που πλήττει και τους έντιμους φορολογουμένους που είναι η συντριπτικότατη πλειοψηφία της κοινωνίας αλλά πλήττει και τα έσοδα των κρατών μελών και τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το θέμα το Κοινοβούλιο θέλει να κάνουμε βήματα και από εγκρίνει εκθέσεις με μεγάλη πλειοψηφία. Η Κομισιόν προτείνει κάποια πράγματα πιο δειλά προς τη θετική κατεύθυνση και πάλι η δυσκολία είναι μέσα στο Συμβούλιο. Επομένως, σας ερωτώ σε έναν ειλικρινή απολογισμό, ποιοι θέλουν και ποιοι δεν θέλουν μέσα στο Συμβούλιο. aitäh äh, Σας ευχαριστώ για αυτά τα ερωτήματα. Όπως σας είπα, η Τραπεζική Ένωση αποτέλεσε μία από τις προτεραιότητες της Εστονικής Προεδρίας ε, και κάναμε μεγάλες προσπάθειες από την πλευρά μας. όπως ήδη ανέφερα κατά την παρουσίασή μου, καταφέραμε να επιτύχουμε πρόοδο σε σχέση με δύο ζητήματα. Πάντοτε στο πλαίσιο της ε, Τραπεζικής Ένωσης, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία σε επίπεδο εκοφή. Αν δείτε τώρα το τι συνέβη στο ΕΚΟΦΗΝ ε, υπήρξαν εκεί διαφορετικές ε, απόψεις από τα κράτη-μέλη αλλά η πλειοψηφία τους ε, θεωρεί ότι καταρχήν θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα της μείωσης του κινδύνου του risk reduction. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το backstop και το σύστημα ασφαλιστικών καταθέσεων. Εγώ προσωπικά ευελπιστώ ότι η Βουλγαρία θα καταφέρει να ολοκληρώσει αυτή τη συζήτηση, αυτή τη διαδικασία, γιατί ήδη έχουν γίνει πολλά, έχουμε εργαστεί εντατικά από αυτού και ήδη η Βουλγαρική Προεδρία έχει θέσει αυτό το ζήτημα προς συζήτηση στο ΕΚΟΦΗΝ του Μαρτίου. Από εκεί και μετά λοιπόν θα δούμε ποια συνέχεια θα μπορέσουμε να δώσουμε στο σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων. Το πρόβλημα είναι ότι βέβαια έχουμε ένα μεγάλο αριθμό κρατών μελών, κατά συνέπεια ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών απόψεων. Ορισμένα κράτη-μέλη ανησυχούν σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και για αυτά τα κράτη-μέλη η αμοιβοποίηση του κινδύνου είναι πολύ πιο σημαντική ενώ για άλλα κράτη-μέλη, για παράδειγμα, προτεραιότητα έχει η μείωση του κινδύνου. Ακριβώς λοιπόν ανάμεσα ε, σε αυτές τις απόψεις θα πρέπει να ε, βρούμε μία χρυσή τομή, να φτάσουμε δηλαδή σε μία συμφωνία, γιατί είναι πολύ σημαντική ομοφωνία σε ό,τι αφορά τα φορολογικά ζητήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μαύρη λίστα. Ναι, υπήρξε εδώ ταχεία πρόοδος Και χαίρομαι που καταφέραμε τελικά στο τέλος της Προεδρίας μας να φτάσουμε εδώ σε μια θέση της πρότασης και σίγουρα εδώ ο στόχος δεν είναι να τιμωρήσουμε κάποια κράτη-μέλη μέσω αυτής της λίστας. Όχι, ο στόχος εδώ είναι να καλέσουμε αυτές τις χώρες, να πιέσουμε αυτές τις χώρες να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαπιστώνω με χαρά μου ότι πράγματι μία σειρά από αυτές τις χώρες ε, επιθυμούν να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν αναλάβει δεσμεύσεις σε υψηλότατο πολιτικό επίπεδο ότι θα προβούν σε μεταρρύθμιση, σε αναθεώρηση των ε, φορολογικών τους οικοδίκων έτσι ώστε να αποφύγουν τη συμπερίληψή τους σε αυτή τη μαύρη λίστα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κίγκολ Ευχαριστώ. Καλωσορίζω τον Υπουργό και θα ήθελα εδώ να θέσω δύο ερωτήματα. Καταρχήν, θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα της μαύρης λίστας των φορολογικών παραδείσων, τη λίστα δηλαδή την οποία προσπαθούμε να καταρτήσουμε τώρα, αλλά γνωρίζετε πως η προσπάθεια αυτή που κάναμε υπονομεύθηκε πολύ γρήγορα γιατί πολλές χώρες συμπεριλήφθηκαν στην γκρίζα λίστα. Από την άλλη, ε, ε, πλευρά βέβαια όπως είπατε θα πρέπει να καλωσορίζουμε τις χώρες εκείνες ε, που κάνουν κάποιες ε, προσπάθειες. Ωστόσο η όλη διαδικασία δεν είναι διαφανής γιατί δεν γνωρίζουμε ποιες χώρες και με ποιον τρόπο έχουν αξιολογηθεί από την ομάδα του κώδικα διοντολογίας ε, του Συμβουλίου. Και κατά συνέπεια δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχουν κάνει αυτές οι χώρες για να περιληφθούν στην κρίτσα λίστα. Οπότε η Εστονία ως μια διαφανής χώρα θα μπορούσε να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και να ταχθεί υπέρ της δημοσιοποίησης ε, των ελόγων ε, αξιολογήσεων και των επιστολών με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι εν λόγω χώρες. Τώρα, από εκεί και μετά είναι ε, ενδιαφέρον το να εξετάζουμε αυτόν τον ε, τις, τις ιστοσελίδες αυτών των φορολογικών ε, παραδείσεων. Ε, μηδενικός, λέμε εδώ, μηδενική επιβολή φόνο σε εταιρείε. Ναι, στην Εστόνια, γιατί έχουμε ε, μηδενικές, τέτοιες, μηδενικούς τέτοιους φόρους σε ό,τι αφορά τα παρακατωμένα κέρδη. Καλώς και αυτό στην Εστονία δεν μας προβληματίζει ιδιαίτερα εφόσον χρησιμοποιείται για ε, τις ε, τοπικές και τις εθνικές δηλαδή ε, επιχειρησιακές δραστηριότητες. Εκείνο όμως που εγώ θα ήθελα να ακούσω είναι ποιος είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων εκείνων που έχουν την έδρα τους στην Εστονία και φορολογούνται στην Εστονία, αλλά των οποίων οι πραγματικοί κάτοχοι, διοκτήτες δηλαδή, βρίσκονται σε άλλες χώρες. Αν λάβουμε μία λίστα από την Εστονία σε σχέση με αυτούς τους πραγματικούς κάτοχους των επιχειρήσεων, τότε θα γνωρίζαμε πραγματικά εάν υπάρχει κατάκτηση, αν δηλαδή ε, λαμβάνει η χώρα φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτά τα ερωτήματα. όταν ε, αναφερόμαστε στο ζήτημα αυτής της λίστας με τις ε, μη συνεργαζόμενες ε, περιοχές δικαιοδοσίας, προφανώς είναι ένα λεπτό ζήτημα. Εμείς υποστηρίζουμε τη διαφάνεια, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με το τι επιθυμούμε εμείς να επιτύχουμε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις επιθυμίες και τα συμφέροντα των χωρών αυτών που θίγονται δηλαδή από την κατάρτιση αυτής της λίστας. Και όπως σας είπα υπήρξαν χώρες οι οποίες ανέλαβαν δεσμεύσεις σε υψηλότατο επίπεδο προκειμένου να μην συμπεριληφθούν σε αυτή τη μαύρη λίστα. Και ακόμα και αν έχουν συμπεριληφθεί στη μαύρη λίστα, εφόσον συμμορφωθούν με ορισμένε προποθέσει, μπορούν να βγουν. Ο στόχος μας εδώ δηλαδή είναι να ενθαρρύνουμε τις τέτοιες χώρες να συνεργαστούν με την Ένωση και όχι να τις φέρουμε σε δύσκολη θέση. Και μπορώ να πω πως σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων οι σχετικές μας ομάδες ε, παρακολουθούν πάρα πολύ προσεκτικά για το κατά πόσο λόγω χώρε πληρώνουν αυτέ τι ε, προποθέσει, αυτέ τι υποχρεώσει ή όχι. Προκειμένου να μην περιληφθούν στη λίστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το φορολογικό σύστημα τη Εστονία, ο κύριο ε, Γκίγκολντ ε, παρεμβαίνει, δεν απαντήσατε στο πρώτο μου ερώτημα. Το πρώτο μου ερώτημα ήταν οι εκθέσει αξιολόγηση και οι επιστολέ με τι δεσμεύσει που ανέλαβαν οι σχετικέ χώρε είναι δυνατόν να δημοσιευτούν. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Σας ευχαριστώ, αλλά ίσως να μην είμαι αρμόδιος για να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Οι είναι εκείνοι μπορούν να του απαντήσουν. Ε, άλλωστε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε σχέση με αυτή τη μαύρη λίστα περιλαμβάνουν μία σειρά από στοιχεία τα οποία ακριβώς εγγυώνται τη διαφάνεια σε σχέση με αυτή τη διαδικασία Εάν θέλετε μπορούμε να εξετάσουμε διεξοδικότερα αυτό το ζήτημα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τους υπόλοιπους ε, συμμετέχοντες στη συζήτηση. Ελπίζω να απάντησα στο ερώτημα σας. Τώρα σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα που θέσατε. Εάν εξετάσετε ευρύτερα το σύστημα, πώς λειτουργεί. Προφανώς ο στόχος των επιχειρήσεων είναι να επιτυχάνουν κέρδη και από εκεί και μετά μέσω μερισμάτων να τα διανέμουν. Εάν δεν θέλουν προφανώς να τα επανεπενδύσουν στην ίδια την επιχείρηση ή να τη διαβρύνουν. Άρα λοιπόν γίνεται η άντληση αυτών των κερδών μέσω μερισμάτων τα οποία διανέμονται και εκεί ακριβώς ε, επιβάλλεται ο φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων. Ναι, προφανώς ε, πριν από ε, δεκαετίες όταν επιβάλαμε σε αυτό το σύστημα στην Αστονία υπήρχαν φόβοι ότι θα ε, οδηγούσαμε τις επιχειρήσεις στην απόκρυψη των κερδών τους αλλά τελικά ε, αυτό δεν συνέβη. Δεν έχω συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για να σας δώσω αυτή τη στιγμή. αλλά και η πραγματική δικαιούχοι που έχουν στην αρρονταπή αξιοποιούν αυτό το σύστημα και κατά συνέπεια είναι υποχρεωμένοι δηλαδή να συμμορφώνονται με το λόγο σύστημα που ισχύει στην Αστονία και δεν έχουμε παρατηρήσει προβλήματα. Μπορείτε να μας τα στείλετε αυτά τα στοιχεία. Ναι, θα στείλετε μια γραπτή ερώτηση, λέει ο Πρόεδρος, και θα σας απαντήσει. Ούτως ή άλλως, όσον αφορά το πρώτο σημείο, το γεγονό ότι όλα τα επιτόκια θα πρέπει, όλα τα συμφέροντα θα πρέπει να προστατεύονται και εκείνη η γνώμη και η εφηβολή του νόμου και το κοινοβούλιο δεν έχει τα ίδια συμφέροντα με τους ανθρώπους που παραβιάζουν τον νόμο. Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Επόμενος ομιλητής για το EFTD δεν βλέπω κάποιον. Η Μπάρμπαρα Κάπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ ε, για την Προεδρία σας, η οποία ήταν επαγγελματική, χωρίς να υπάρξουν εκνευρισμοί, πράγμα το οποίο προφανώς είναι επιθυμητό. Ε, και όπως είπατε και εσείς στην παρουσίασή σας, αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε μια, διερχόμαστε μια θετική τάση σε ό,τι αφορά δηλαδή την, ε, το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, αλλά και τα όσα σύνουσες με το εργατικό δυναμικό. Επίσης ε, σωστά είπατε ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ακριβώς αυτόν την, ε, την ε, όθηση της ανάπτυξης προκειμένου να προβούμε στην, σε αυτές τις, στα νέα συστήματα, στην εδρίωση των νέων συστημάτων και σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου Πράγματι είναι σημαντικό αυτό να γίνει, όπω αναφέρθηκε ήδη, αλλά αναφερθήκατε βέβαια και στην, ε, στην ψηφιακή οικονομία, στον χώρο τη ε, χρηματοοικονομική δραστηριότητα, ε, αλλά και στο πλαίσιο των τραπεζικών υπηρεσιών, των πληρωμών δηλαδή των ψηφιακών. Ενώ αναφερθήκατε βέβαια και στο e-residency πρόγραμμα της Εστονίας, όπου υπάρχει δηλαδή ένα ψηφιακό footprint, αν θέλετε, του κάθε πολίτη. Τρία όμως ζητήματα κατά τη δική μου άποψη δεν επιλύθηκαν στο πλαίσιο της δικής σας Προεδρία. Καταρχήν το πακέτο για τις υπηρεσίες, στο πλαίσιο του οποίου το e-residency θα μπορούσε να έχει αποτελέσει μια βέλτιση πρακτική σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του. Μετά, ε, τις διατάξεις ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τι ηλεκτρονικέ δημοσιεύσει και τα e-books δεν φτάσαμε σε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά δηλαδή την επιβολή ενό μειωμένου φορολογικού συντελεστή. Ε, και από εκεί και μετά η ε, τα όσα προβλέπουμε σε ό,τι αφορά την επιβολή, ε, επιβολή τελών για τους διαμεσολαβητές και πάλι δεν επιτύχαμε μία πρόοδο. Αυτοί οι τρεις φάκελοι μαζί με κάποιου φακέλου από το βιομηχανικό τομέα, για παράδειγμα, διατάξει ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων σε σχέση με τι ηλεκτρονικέ επικοινωνίε, η οδηγία σε ό,τι αφορά ε, την, ε, τα δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησία, ε, περνάνε τώρα στα χέρια της Βουλγαρικής Προεδρίας. Εσείς λοιπόν τι συμβουλή θα είχατε να, δώσει στην, ε, να δώσετε στην Βουλγαρική Προεδρία σε ό,τι αφορά την πρώτη που θα μπορούσε να επιτύχει στον ψηφιακό τομέα. Ένα δεύτερο ερώτημα τώρα. Αυτή η λίστα των μη συνεργαζόμενων ε, περιοχών δικαιοδοσίας, των χωρών δηλαδή που αναφέρθηκαν επανειλημμένα. Ε, ένα μεγάλο επίτευγμα της δικής σας Προεδρίας ήταν ακριβώς το πρώτο βήμα που επιτύχατε σε ό,τι αφορά την κατάρτιση αυτής της μαύρης λίστας. Το γεγονός όμως ότι τώρα μέσα σε ένα μήνα ήδη 8 χώρες βγήκαν από αυτή τη λίστα παρά το σεβασμό που σας τρέφουμε και παρά τη διαφάνεια που υπήρξε στη διαδικασία δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς τόσο γρήγορα βγήκαν αυτές τις χώρες. Οπότε θα θέλαμε να σας εξηγήσετε καλύτερα πώς ακριβώς έγινε αυτό, γιατί βγήκαν αυτές τις χώρες από τη λίστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Όσον αφορά τους ε, δεσμευτικούς κανόνες ε, για τους ε, διαμεσολαβητές και τους φορολογικούς συμβούλους, η πρόταση δημοσιεύθηκε αμέσως πριν την έναρξη της Προεδρίας μας. Πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη πρόταση. Χρειάζεται εις βάθος συζήτηση πολλών ζητημάτων και συζητήθηκε η πρόταση σε πολλές συνεδριάσεις και καταλήξαμε σε δύο συμβιβαστικές προτάσεις, αλλά όπως γνωρίζετε η Προεδρία έξι μήνες διαρκεί. Επομένως δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στα τελικά συμπεράσματα. Πιστεύω ότι η πρόταση είναι έτοιμη για την επόμενη Προεδρία, η Βουλγαρία δηλαδή, μπορεί να προχωρήσει και να οριστικοποιήσει το αποτέλεσμα. Όσον αφορά τους κανόνες ΦΠΑ, η ε, φορολογία των ηλεκτρονικών βιβλίων και των ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων δυστυχώς αυτό είναι ένα από τα θέματα στα οποία ε, δύο κράτη-μέλη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία και επειδή χρειάζεται ομοφωνία για το θέμα αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ε, το είδαμε και στη διάρκεια της Μαλτέζικης Προεδρίας. Προσπάθησαν να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία και δυστυχώς ούτε και εμείς καταφέραμε να έχουμε κάποια πρόοδο στο θέμα αυτό. Για την ερώτησή σας για τη μαύρη λίστα. Πράγματι, αφενός ε, θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι το γεγονός ότι έχουν αφαιρεθεί ήδη 8 χώρες από τη μαύρη λίστα αποτελεί αδυναμία, αλλά μπορεί να αποτελεί και το δυνατό μας χαρτί, διότι το γεγονός ότι υπάρχουν ε, χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, επειδή φοβούνται ότι θα καταλήξουν στη μαύρη λίστα ή έχουν ήδη βρεθεί στη μαύρη λίστα, έχουν λάβει ε, σοβαρά μέτρα για να αλλάξουν την νομοθεσία τους και να ε, μπορέσουν να αφαιρεθούν από τη λίστα, είναι θετικό. Ο κύριος Νέντερμαϊερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την Εστονία για μια πάρα πολύ καλή προεδρία. Μία ερώτηση έχω μόνο όσον αφορά μια πολύ ουσιαστική πρόταση, την, ε, το CCTB, την κοινή φορολογική βάση επιχειρήσεων. Ε, ξέρω ότι υπάρχουν ε, περίπλοκα θέματα και δεν μπορεί κανείς να περιμένει να λυθούν τα θέματα αυτά στη διάρκεια μιας προεδρίας, αλλά θα ήθελα να ακούσω πρώτον την προσωπική σας άποψη και δεύτερον και μια πρόβλεψη. Πώς βλέπετε να προχωρά το θέμα αυτό τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Πράγματι, στη διάρκεια της Εστονικής Προεδρίας ασχολήθηκαμε με την πρόταση για το CCTB. Ε, έγινε η πρώτη ανάγνωση και ολοκληρώθηκε και η κατάρθρο εξέταση ε, στα κεφάλαια 1 5. Ταυτόχρονα ξεκίνησαν και συζητήσεις για τη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας, κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με την πρόταση για την κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων. Εκεί υπήρξαν συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις ε, εναλλακτικές λύσεις ε, για τον τομέα της φορολογίας της ψηφιακής οικονομίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το ζήτημα αυτό και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Ε, υπάρχουν διεστάμενες απόψεις μεταξύ των κρατών μελών. Προσωπικά φρονώ ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για το θέμα αυτό, αλλά βεβαίως η προσωπική μου άποψη δεν έχει καμία σημασία στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ, ο κύριος Φερνάνδες. Ευχαριστώ πολύ. Να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου την Προεδρία και θα ήθελα και πάλι να αναφερθώ στις διαπραγματεύσεις ε, για την πρόοδο για την ε, Τραπεζική Ένωση. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει μια επίφαση συζήτησης ε, για τα μέτρα για την μείωση των κινδύνων και τα μέτρα για την αμοιβοποίηση των κινδύνων. Διότι συζητήσεις ε, ε, όπως η οδηγία δεν είναι πρόταση μόνο για αμοιβοποίηση αλλά είναι και πρόταση για μείωση των Και αυτό που προσπαθούμε να καταφέρουμε στην Ένωση, στην, Ευρωπαϊκή, ε, στην Ευρωζώνη, είναι να μειώσουμε τους κινδύνους. Και το ε, είναι πρόταση για να μειώσουμε τους κινδύνους. Εσείς είπατε ότι υπήρξε πρόοδος, ιδίω όσον αφορά το θέμα της μείωσης των κινδύνων. Νομίζω ότι και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο προχωρούν με τον κανονισμό, αλλά όπως έλεγε και ο συνάδελφος ο κ. Παπαδημούλης, η πρόοδος είναι ισχνότατη. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς ε, διεμήφθη η συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο. Ξέρουμε ότι ακόμα δεν έχει περάσει σε πολιτικό επίπεδο το θέμα, αλλά θα ήθελα κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για τη συζήτηση στο τεχνικό επίπεδο και να επιμείνω και πάλι ε, στο εξή. Τι προβλήματα υπάρχουν, ποιε χώρε είναι αυτέ οι οποίε μπλοκάρουν και πώ μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε το ζήτημα στη διάρκεια τη παρούσα Προεδρία που ξεκινάει τώρα. Νομίζω ότι οι διαιρέσει που όπω έλεγα και πριν μεταξύ τη μείωση και τη αμοιβοποίηση είναι στρεβλή. Όλα ουσιαστικά αποτελούν θέμα μείωση του κινδύνου και θα ήθελα να μα πείτε κάποιε περισσότερε λεπτομέρειε για την πρόοδο για τη συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Όπως είπα ήδη, για την Τραπεζική Ένωση η Τραπεζική Ένωση αποτέλεσε ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα που απασχόλησαν την Εστονική Προεδρία και αφιερώσαμε και ε, χρόνο και πόρους ε, στη συζήτηση για το θέμα αυτό. Οι συνεχίστηκαν σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ και νομίζω ότι ακόμα και τώρα είναι σαφές ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των κρατών μελών επί του θέματος. Κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ότι η αμοιβοποίηση του κινδύνου είναι το πιο σημαντικό και είναι ο πιο σημαντικός τρόπος να προχωρήσουμε και κάποιες άλλες χώρες θεωρούν ότι πρώτα πρέπει να μειωθούν οι κίνδυνοι και μετά να γίνει η αμοιβοποίηση και να προχωρήσουμε όσον αφορά τις τεχνικές εργασίες ε, για το πρόγραμμα της ε, εγγύησης των καταθέσεων, ε, οι προτεραιότητες ήταν για μεθόδους μείωσης των κινδύνων. Όπως ξέρουμε το θέμα αυτό έχει προχωρήσει καλά και η Εστονία προχώρησε τον οδικό χάρτη που είχε συμφωνηθεί το 2016 με τα χαράς δεν να σας πω ότι καταρρίξαμε και σε κάποιο συμπέρασμα με το Κοινοβούλιο όσον αφορά την βαθμολογία των ε, μη ασφαλών προϊόντων και το θέμα για τις μεταβατικές διατάξεις ε, για το ε, ε, IFRS. Τώρα, τα προβλήματα εξαρτώνται από το, ε, την άποψη ποια χώρα θεωρούμε ως βάση. Όπως σας είπα υπάρχουν κάποιες χώρες ε, σκανδιναβικές ή πιο συντηρητικές χώρες ε, που έχουν μία άποψη και οι νότιες χώρες θεωρούν ίσως ότι η αμοιβοποίηση είναι η κατάλληλη επιλογή. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε κάποιο συμβιβασμό επ' αυτού, αλλά σε τεχνικό επίπεδο, παρά τις σκληρές μας προσπάθειες και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάγκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που είστε εδώ και να σας συγχαρώ και για την πρόοδο που έχετε επιτύχει στην Προεδρία σας. Την εκτιμούμε ιδιαίτερα, δεδομένου ότι γνωρίζω ότι η Εστονική Προεδρία δούλεψε και πολύ στο περιθώριο ε, για τα δύσκολα θέματα, κυρίως για την κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων και ξέρω ότι η φορολογία είναι ακαθόδε ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, με χαρά άκουσα και την προσωπική σας άποψη ε, που είπατε ότι πιστεύετε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία βλέπουμε ότι και η νέα γερμανική κυβέρνηση που είναι ακόμα υποσύνθεση ε, υποστηρίζει ε, να υπάρχει μια ευρωπαϊκή φορολογική βάση και να ελάχιστο, ε, και ένας ελάχιστο φορολογική συντελεστής. σε ποιο σημείο πιστεύετε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι εξή. είδατε και τι δυναμικές υπάρχουν όσον αφορά την φορολογία. Δέκα χώρες προσυπογράφουν ε, την επιστολή την οποία ξεκίνησε ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών ο Μπρουνολεμέρ. Πιστεύετε κι εσείς ότι μπορούμε να υπερκεράσουμε τις διαφορές σε σύντομο χρονικό διάστημα και ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει τα ενία. Είναι περισσότερο πολιτική ερώτηση. Θα πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει τα ενία στη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας, να μην περιμένουμε τον ΩΣΑ, να μην περιμένουμε την Αμερική να δράσει, αλλά να ξεκινήσουμε εμείς πρώτοι. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η Εστονία έκανε πολύ κόπο για το θέμα της ε, κοινή ε, φορολογικής βάσης των επιχειρήσεων. Δεν θα αρχίσω τώρα να σας λέω πού καταλήξαμε στη συμφωνία και πού όχι, διότι στη διάρκεια της Προεδρίας μας σε κάποιες χώρες μέλη είχαμε εκλογέ. Και αυτό φυσικά πάντα δυσχεραίνει περισσότερο την επίτευξη συμφωνίας. Οι νέες κυβερνήσεις, συνασπισμοί, ενεξελίξεις σημαίνει ότι οι υπουργοί στην πραγματικότητα δεν έχουν ακόμα εντολές και δεν είναι απαραίτητος κατά, αλλά δεν μπορούν να λάβουν θέση. Και αυτός είναι και ο λόγος ε, που κάποιες πιθανές συμφωνίες ε, καθυστέρησαν περισσότερο από ό,τι φανταζόμασταν. Φορολογία της ψηφιακής οικονομίας, σαφώς ε, σημαντικό ζήτημα. Στην Ευρώπη έχουμε θέσει το θέμα στο θεματολογιό μας και ακριβώς ε, επειδή η Ευρώπη ήταν αυτή που το έθεσε, ο ΣΑ πλέον πιέζεται. Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένες φορές δεν αντιλαμβάνονται ότι η καλύτερη λύση θα ήταν ε, μια παγκόσμια συμφωνία για φορολόγηση. Είμαι υπέρ της πρωτοβουλίας ε, των κρατών μελών ε, που επιθυμούν ε, να προχωρήσει η διαδικασία πιο γρήγορα. Αυτή είναι πράγματι μία από τις πιθανές εναλλακτικέ λύσεις. Και σε αυτή την περίπτωση σίγουρα προτιμούμε να υπάρχει κοινή δράση από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό φυσικά μέχρι να καταλήξουμε σε μια διεθνή συμφωνία για το πώς θα πρέπει να φορολογείται η ψηφιακή οικονομία παγκοσμίω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαυρίδης, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Right oh, um, εγώ θα ξεκινήσω με μια ερώτηση που αφορά τους κοινωνικούς δείχτες, οι οποίοι ήταν και το κύριο, ένα από τα κύρια θέματα στο Γκέντερμποκ της Σουηδίας. Εκεί υπήρξε η θέση ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν οι κοινωνικοί δείχτες ή ένα μέρος τους στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Θα ήθελα να ξακούσω την θέση σας πάνω σε αυτό το θέμα. Και το δεύτερο θα επαναφέρω στη συζήτηση το καυτό θέμα με το ήτης. αλλά από την ανάποδη πλευρά. Σας είχα, παρακολουθήσει προσεκτικά στην εισαγωγή σας, στην αρχική σας εισαγωγή και μιλήσατε για sufficient progress on the European Banking Union. Θα συμφωνήσουμε. Πράγματι υπήρξε σημαντική πρόοδος εφαρμόστηκαν οι δύο πρώτοι πυλώνες. Έχουμε μηχανισμούς στήριξης και χρηματοδότησης των τραπεζών. Έχουμε την οδηγία για την εξυγίαση των τραπεζών. Με αυτά δεν είναι εύλογο να διαρωτηθεί κάποιος τι είναι οι πραγματικοί λόγοι και όχι οι τεχνικοί που προβάλλονται. Οι πραγματικοί λόγοι για τον οποίο δεν προχωράμε στον τρίτο πυλώνα ο οποίος ήταν εξ αρχής αναπόσπαστο μέρος του European, του European Banking Union. Γιατί αν θέλαμε ο καθένας μας να προβάλλει τεχνικούς λόγους, θα, θα μπορούσαμε να τους προβάλλουμε και για τον πυλώνα τον πρώτο και για τον πυλώνα τον δεύτερο. Θα ήθελα λοιπόν από εσάς μια ειλικρινή εκτίμηση γιατί δεν προχωράμε παρακάτω. Αυτό είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους μας, γιατί η υποψία, μας είναι να μην τρέχουμε εκ των υστέρων για προβλήματα που θα δημιουργηθούν γύρω από τον τραπεζικό τομέα. Σας ευχαριστώ. Äh, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση και να σας πω πως για το πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει με τους κοινωνικούς δείκτες και το Γκέτεμπουργκ και το κατά πόσο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, να σας πω τα εξή. Εμείς πρέπει να δούμε την όλη διαδικασία και να τη δούμε ε, σαν κάτι το οποίο είναι ένα σύνολο. Έχει βελτιωθεί το εξάμεινο, είναι πιο στοχευμένες οι συστάσεις. Αληθεύει βέβαια το ότι δεν έχουμε καλύψει όλες τις προσδοκούμενες, όλους τους προσδοκούμενους στόχους ε, και πως η αναχώραση στάσεις θα μπορούσαν να είναι καλύτερες, αλλά ναι, κατανοώ αυτό που λέτε και οι κοινωνικοί δείκτες έχουν ένα ρόλο να παίξουν μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να αναλύσω το μέγεθος που θα πρέπει να έχουν αυτοί οι δείκτες και δεν μπορώ καν να σας πω πόσο έχουμε προχωρήσει σε σχέση με τις αρχές που συζητούσαμε στο Γκέτεμπουργκ. Τώρα για τον τρίτο πυλώνα και για το θέμα του συστήματος εγγύησης καταθέσεων, είναι τόσα πολλά τα κράτη-μέλη που κάθονται στο τραπέζι. Και κάθε κράτος μέλος και κάθε κυβέρνηση έχει το δικό της εκλογικό σώμα με τα δικά του προβλήματα. Και θα πρέπει να βρούμε κάποιο είδους συνένεση. Οπότε η δική μου εντύπωση είναι πως ναι, συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σταδιακά, βήμα-βήμα, θα ξεκινήσουμε με τη μείωση κινδύνου και μετά, παράλληλα μάλλον, θα συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα βήματα. Αλλά αν προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα, τότε τελικά δεν θα φτάσουμε πουθενά. Αυτή είναι η δική μου άποψη. και είμαι βέβαιος πως με τον τρόπο αυτό θα καταλήξουμε σε συμφωνία και στο θέμα αυτό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων. Ευχαριστώ πολύ και εγώ ελπίζω πως θα συμβεί κάτι τέτοιο και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, για την εξαιρετική αυτή ανταλλαγή απόψεων και καταγράφω πως όλες οι πολιτικές ομάδες συνεχάρισαν την Προεδρία της Εστονίας και θα ήθελα απλώς να επαναλάβω και εγώ το ότι η αξιολόγηση που γίνεται της Προεδρίας σας ήταν πολύ πετυχημένη και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας μια και παραμένετε υπουργό του ΕΚΟΦΗΝ. Και ελπίζω πως αυτή η καλή συνεργασία θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μερικέ ανακοινώσει που πρέπει να κάνουμε στα γρήγορα πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, την οποία έχουμε εγκρίνει. Και να σας πω, τις 14 Δεκεμβρίου συντονιστές αποφάσεις αναβάλαμε ε, το θέμα του πακέτου για την νομισματική ένωση όχι για την νομισματική ένωση για το ΦΠΑ ναι για το πακέτο για το ΦΠΑ να σας πω πως Χτες ε, διορίσαμε και θα τα δείτε την επόμενη φορά. Λοιπόν, όλα για τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε τώρα. Να σας πω για την αποστολή στην Αθήνα πριν το καλοκαίρι και επίσης το πρόγραμμα της χώρας θα αξιολογηθεί, ανταγωνισμός εγκρίθηκε Έχουμε και το, τη μόνιμη ε, ομάδα. Τα υπόλοιπα πρέπει να σας πω ότι ψάχνουμε να βρούμε για τις τρεις πρώτες συναντήσεις ε, τις κατάλληλες ημερομηνίε. Σύσταση αποστολής Γαλλία, ΕΛΚ. Τρία για, το, ε, για ε, δύο ε, ένας από Άλτε και ένας από Πράσινους και να σας πω πως για τα υπόλοιπα θα ενημερωθείτε και για τους υπόλοιπους ε, θα τα βρείτε γραπτά. Να σας πω πως ε, θα πρέπει να βρούμε και συνάντηση για να συναντηθούμε με τον Μάριο Σεντένο που θα γίνει αφού αναλάβει η καθήκοντα και με τον νέο γραμματέα και επίσης για την στατιστική γνωμοδοτική υπηρεσία καλέσαμε προτάσεις από τους συντονιστές. Θα ψηφίσουμε σήμερα για το διορισμό, οικονομική διακυβέρνηση, ημερομηνίες. Εκεί εγκριθήκαν στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής εβδομάδας. Follow-up, πακέτο της Κομισιόν για την ΟΝΕ. Εκατεξιοδότηση πράξη και άλλες εφαρμοστικές πράξεις. Συντονιστές θα κάνουν προτάσεις ε, για την ε, συνάντηση του Φεβρουαρίου, γραπτά. Δημόσια ακρόαση μέσω θα αποφασίσουν οι συντονιστές για το θέμα ε, των χρηματοπιστωτικών. Brexit συντονιστές συζητάνε τη μεθοδολογία εργασίας. Ψήφισμα αποφασίσαμε το σχετικό ψήφισμα να μην δώσουμε συνέχεια. Για το ελεγκτικό συνέδριο, συντονιστές να υποβάλουν προτάσεις για θέματα προτεραιότητας για το πρόγραμμα εργασίας αυτών για το 19 ασφαλής και αντασφαλίσεις ημερομηνία τροπολογίας 14 Δεκεμβρίου καμία τροπολογία δεν κατατέθηκε Δεν θα συζητηθούν λοιπόν, κατευθείαν θα ψηφίσουμε για το σχέδιο γνωμοδότησης. Αυτά. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Η ημερομηνία της εφαρμογής για τα θέματα μεταγραφής Στο ψήφισμά μας ζητήσαμε μία αναβολή της θέσης σε ισχύ για το IDD και εκεί μεγάλη πλειοψηφία ε, το δέχτηκε. Γίνεται και κάποια, κάποιο συντονισμός με το Συμβούλιο έτσι ώστε να είμαστε ως τον ταχύτεροι. Μας είπε ποιες τροπολογίες θέλει. Λογικά όλα αυτά. μια πλουστευμένη διαδικασία του 52 μας επιτρέπει να σεβαστούμε σχετικά τις καταληκτικές προθεσμίες. Θα τα πούν οι εισηγητές. Ο Βέρνερ λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. από άποψη σε χρονικής συγκυρία, η διαδικασία είναι πολύ δύσκολη, οπότε θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εσάς προσωπικά πρόεδρε Θερμά και την Γραμματεία για το γεγονός ότι προετοιμάσατε με τέτοιο τρόπο τις εργασίες μας έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να παρατείνουμε τις σχετικές ημερομηνίε. Τώρα, ε, το γεγονός ότι η Επιτροπή έλαβε τη σχετική απόφαση τόσο καθυστερημένα τόσο σε ό,τι αφορά τον κατεξοδότηση κανονισμού αλλά και σε ό,τι αφορά τον, την οδηγία δεν οφείλεται στις καθυστερήσεις από την πλευρά του εισηγητή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά στην, ε, στο μηχανισμό που έχει προβλέψει τις αποφάσεις της ίδια η Επιτροπή. Η Επιτροπή δηλαδή ήθελε να, να, να υποβάλει τι σχετικέ προτάσει ε, πριν από το ε, θερινό διάλειμμα. Μετά καθυστέρησε πολύ μετά από το θερινό διάλειμμα να τις υποβάλει. Και από εκεί και μετά οι προτάσει τροποποίησης που κάναμε εμείς ε, Κατά συνέπεια, σε ό,τι αφορά το ίδιο το κείμενο τη οδηγία, ήρθαν πολύ καθυστερημένα με τη σειρά του. Τώρα, καταρχήν, επιτρέψτε μου να πω κάτι σε ό,τι αφορά την κατεξουδότηση πράξη. Εδώ έχουμε ε, προτείνει να μην υπάρξει αντίρρηση από δική μα πλευρά και ούτε υποβλήθηκαν τροπολογίε από συναδέλφου. Οπότε αύριο το πρωί θα μπορέσουμε να προβούμε στην ψηφοφορία χωρί κανένα πρόβλημα. Δύο παράγραφοι είναι αυτέ που μα αφορούν. έξι αιτιολογικές σκέψεις και έξι περαιτέρω αναφορές μέσα στο κείμενο, ε, επί των οποίων θα ψηφίσουμε αύριο. Ποιο είναι το, το, το, η κεντρική ιδέα, αν θέλετε, αυτών των αλλαγών, τόσο στην οδηγία όσο και την εξοδότηση κανονισμού η μεταφορά ουσιαστικά τη ημερομηνία σε θέση σε ισχύ ή μάλλον εφαρμογή ε, του κανονισμού και ε, των κατεξοδότων του κανονισμού από τι 23 Φεβρουαρίου στην 1η Οκτωβρίου. Γιατί είχαμε συμφωνήσει ότι πράγματι είναι υπερβολικά βραχή το χρονικό διάστημα για την εφαρμογή ε, του κανονισμού στα κράτη-μέλη. Και επειδή αποφασίσαμε να μην υπάρξει αναβολή της μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία, απλώς ε, αποφασίσαμε να μετατεθεί ουσιαστικά η εφαρμογή, υποχρέωση εφαρμογή αυτών των νέων διατάξεων από τον κλάδο τον Οκτώβριο του 2018. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε στο Συμβούλιο, τα 15 από 28 κράτη-μέλη αξίωσαν την παράταση της μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία δηλαδή και ε, την, ε, ημερομηνία μεταφοράς ε, της, στην Εθνική Νομοθεσία από τις 23 Φεβρουαρίου στην 1η Ιουλίου του 2018. Ε, παρότι δύο μεγαλύτερα κράτη-μέλη, η Γαλλία και η Γερμανία, δεν συμφώνησαν με αυτή την πρόταση, εγώ θεωρώ πω ε, θα είχε νόημα μια τέτοια παράταση. Για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και άλλα κράτη-μέλη θεώρησαν πω θα ήταν σκόπιμη μια τέτοια ε, παράταση τη ε, μεταφορά στην εθνική νομοθεσία και κατά συνέπεια έναρξη ισχύω. Αλλά κάτι τέτοιο βέβαιο, βέβαια θα προπέθεται μια πρόταση ε, από την πλευρά τη Επιτροπή για τροποποίηση του κειμένου τη ίδια τη οδηγία. Η εν λόγω πρόταση υποβλήθηκε και αυτή καθυστερημένα από την Επιτροπή, συγκεκριμένα στι 23 ε, Δεκεμβρίου. Ε, και βέβαια δεν είχαμε κάποια άλλη ε, συνεδρία στη δική μας, της Επιτροπής μας πριν από το ε, διάλειμμα για τα ε, Χριστούγεννα γιατί αν το είχε υποβάλει, αν είχε υποβάλει την πρόταση της μία εβδομάδα νωρίτερα Επιτροπή θα είχαμε αποφύγει όλες αυτές τις καθυστερήσεις, όλα θα είχαν γίνει εντός των προθεσμιών αλλά εν τη σοφία της Επιτροπή αποφάσισε τότε να υποβάλει την πρότασή της. Τώρα, τι μας προτείνει σε αυτήν τη νέα πρόταση. Ουσιαστικά τροποποίηση της, ε, της προβλεπόμενης ε, μεταφοράς ε, στην Εθνική Νομοθεσία και εφαρμογής και θέση ισχύ στην 1η Ιουλίου του 18 σε ό,τι αφορά τους δύο κανονισμούς 1η Οκτωβρίου του 18 και μετά στο δεύτερο άρθρο αναφέρεται και είναι σημαντικό θα ισχύει με αναδρομική ισχύ από τις 23 Φεβρουαρίου του 2018. Ουσιαστικά δηλαδή η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ με αναδρομική ισχύ αναδρομική ισχύ σε ό,τι αφορά τι 23 Φεβρουαρίου του 2018. Και γιατί κάτι τέτοιο είναι σημαντικό, γιατί ανάμεσα στην επόμενη ολομέλειά μας και τον Ιουλίου, σε αυτό το ενδιάμεσο διάστημα, θα πρέπει να υπάρξει και ένα διάλειμμα στο πλαίσιο του διαλόγου που θα γίνει ε, μεταξύ ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Άρα λοιπόν ε, σε αυτό το, σε αυτό το, μέσα σε αυτή την προθεσμία ε, θα, ουσιαστικά θα προκύψουν από τις 23 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου ε, μία εβδομάδα θα προσύψει ε, νομικού κενού αν θέλετε γι' αυτό έγινε αυτή η πρόταση από την ε, ε Επιτροπή τη αναδρομική ισχύω, δηλαδή από τι 23 Φεβρουαρίου, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα ασφαλείας δικαίου σε ό,τι αφορά την λόγο περίοδο. Αυτή είναι λοιπόν η πρόταση που μα υπέβαλε η Επιτροπή και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει από του συναδέλφου θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στην ψηφοφορία ε, την αυριανή και αυτό το ζήτημα και αυτή την πρόταση έτσι ώστε να μπορέσουμε την ερχόμενη εβδομάδα να αποφασίσουμε επισήμω πλέον σε επίπεδο και να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε λοιπόν και τι ε, ε, σχετικές τροποποίησεις των κατοξιδότησης και ε, της ε, οδηγίας που ουσιαστικά αφορούν, όπως είπαμε, μόνο αλλαγή ημερομηνιών. Από εκεί και μετά, εγώ ε, έκανα και μια συζήτηση με τον ε, Βούλγαρο ακόλουθο για θέματα οικονομικών, ο οποίος μου διαβεβαίωσε ότι πράγματι θα ε, ολοκληρώσει θετικές συζητήσεις σε επίπεδο Συμβουλίου εγκαίρως, έτσι ώστε πραγματικά δηλαδή να υπάρξει και από τις δύο πλευρές η σύμφωνη γνώμη. Σα ευχαριστώ εκ των προτέρων για την υποστήριξή σα, συνάδελφοι, και πραγματικά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε αυτή την πρόταση χωρί ιδιαίτερα προβλήματα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λάγκη. Προσπαθήσατε να λύσετε ένα πολύ περίπλοκο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν προέκυψε από δικό μας φάλμα, αλλά νομίζω ότι το Κοινοβούλιο με πολύ ευφύ τρόπο προτείνει μια λύση. και εκπροσωπώντας και την ομάδα μου πολύ σωστά περιγράψατε την τροπολογία που ζήτησε το Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε πλήρη ευθυγράμμιση γιατί διαφορετικά δεν θα σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την διατύπωση που προσθέθηκε που ήταν το at the latest για να δούμε αν κάποιοι μπορούν να προχωρήσουν ε, αφού είναι έτοιμοι. Λύθηκε λοιπόν το πρόβλημα και αυτή τη στιγμή στηρίζει όλες τις προτάσεις το Συμβούλιο. Πλήρης ευθυγράμμιση λοιπόν μεταξύ των συνομοθετών. Και σας ευχαριστώ γιατί αυτή η διάταξη για την αναδρομική ισχύ θα λήξει και το πρόβλημα των λίγων ημερών όπου δεν θα προλάβουμε τις ημερομηνίες. Και αν μα είχε δώσει η Κομισιόν το κείμενο μια εβδομάδα νωρίτερα δεν θα είχαμε το πρόβλημα. Αυτό εν πάση περιπτώσει του ευχαριστούμε. Ξέρουμε πως ήταν ε, δύσκολο το θέμα στα διάφορους ορόφους του κτηρίου. Χρειάστηκε να περιμένουμε να κατέβει τις σκάλες, να πάρει το ασανσέρ, ο φάκελος και να φτάσει μπροστά μας. να δώσουμε μία λέξη, με μία λέξη σαφήνεια στους, στις αγορές. Αύριο θα ψηφίσουμε. Συγγνώμη, σήμερα το απόγευμα θα ε, ψηφίσουμε για τα θέματα τα υπόλοιπα που υπάρχουν αντιρρήσει και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία του 52. Οπότε, ο εισηγητής διατυπώνει τροπολογίες παρόμοιες, πανομοιότυπες με αυτές του Συμβουλίου και δεν χρειάζεται τριμερίς γιατί είναι πανομοιότυπα τα κείμενα. Και μετά έχουμε τις 7 εβδομάδες για τη δυνατότητα ενστάσεων και μετά αυτομάτως υιοθετείται το κείμενο. Οπότε δεν θα γίνει τριμερής και θα είναι στην επίσημη εφημερίδα λίγες μέρες μετά την προθεσμία το κείμενο, οπότε κανένα πρόβλημα. Στηρίζω λοιπόν τις προτάσεις του εισηγητή, του Συμβουλίου. Και θα σας στηρίξουμε και στην ψηφοφορία που θα γίνει αργότερα σήμερα. Έτσι είμαστε και ρεαλιστές. Η Ευρώπη καμιά φορά έχει τη δυνατότητα να σπεύσει. Δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος, μετά τους Σκιώδης. Και καλωσορίζω βέβαια Ashley Fox, Sophie De Welt. Πού είναι οι Σκιώδης. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, τον κύριο Λάγκερ, και για τα λόγια του και για τη στήριξη που προσφέρει. Εμείς προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε τις συστάσεις και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή ε, του θέματος αυτού, του IDD, και κατανοήσαμε πως κάποιες, κάποιες από τις ασφαλιστικές και κυρίως οι μισέου μεγέθους θα ήθελαν να δείξουμε κατανόηση γιατί έχουν τεχνικές δυσκολίες ε, με την εφαρμογή της οδηγίας και γι' αυτό προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε τις αισθάνσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά Είχαμε τεχνικές ε, δυσκολίες με το πρόγραμμα και γι' αυτό η πρόταση αυτή εγκρίθηκε μια, μια μικρή καθυστέρηση. Καταγράφουμε τώρα τις θέσεις κάποιων μελών του Συμβουλίου. Καταγράφουμε την επιστολή που έστειλε η ΕΚΟΝ σε εμάς και ελπίζουμε πως θα καταφέρουμε να βρούμε μια ρεαλιστική ε, λύση που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Βέρνα, θέλεις να απλήσεις κάποια συμπεράσματα τη συζήτηση. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη και επαναλαμβάνω ότι χωρίς την υποστήριξη του Προέδρου και της Γραμματείας της Επιτροπής ΕΚΟΝ εδώ δεν θα είχαμε καταφέρει να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία, η οποία μα επιτρέπει τελικά να επιτύχουμε περισσότερη ασφάλεια δικαίου. Ναι, και πράγματι, Πρόεδρε, αν είναι απαραίτητο ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα, όχι. Αρνητικό νεύμα από την ε, γραμματεία. Α, δεν θα ψηφίσουμε καν από αυτού. Καλώ, ακόμα καλύτερα. Πρόεδρος. Θα αξιοποιήσουμε τη διαδικασία του 52, με βάση την οποία θα μας παρουσιάσετε το κείμενο και από εκεί και μετά αυτό θα υιοθετηθεί αυτομάτως εκτός και αν εκφραστεί αντίρρηση από ένα απαραίτητο αριθμό είτε μελών είτε πολιτικών ομάδων, δηλαδή ένα απαραίτητο κατόφλι. Καλώς, αυτή τη διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα Okay. Καλώς. Θα διακόψουμε για 5 λεπτά.

Dear Ας ξεκινήσουμε συνάδελφοι. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ τον Υπουργό, Οικονομικών της Βουλγαρίας και Πρόεδρο του ΕΚΟΦΕΝ, τον κύριο Βλάντισλαβ Γκόρανοφ. Τον ευχαριστώ για την παρουσία του σήμερα εδώ. Το Γιονός, ε, ότι αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας για να μας παρουσιάσει σήμερα εδώ τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής ε, Προεδρίας στον τομέα βέβαια των οικονομικών ήδη συνεργαζόμαστε στενά με την Προεδρία σας και ε, σας συγχαίρω ήδη για το πρόγραμμα εργασιών σας και για τη συνεργασία που έχετε ξεκινήσει ήδη με την Επιτροπή μας. με βέβαιος ότι θα έχουμε μια οικοδομητική συνεργασία. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία για την Προεδρία σας, καθώς η επιτυχία της δικής σας Προεδρία θα αποτελέσει και επιτυχία δική μας. Γιατί βέβαια στο πλαίσιο αυτού εδώ του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα εξεταστούν μία σειρά από κέρια σημασία σε φάκελο, οπότε θα πρέπει να φτάσετε σε συμφωνία επί μία σειρά θεμάτων, θα ξεκινήσουν τριμερείς διάλογοι για κάποια από αυτά, οπότε θα πρέπει να συνεργαστούμε εύρυθμα μεταξύ μας και νομίζω πως ε, ήδη ξεκινήσαμε πολύ καλά. Συζητήσαμε δηλαδή μόλις τώρα ε, και ε, την οδηγία σε ό,τι αφορά τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων και καταλήξαμε στο ότι θα μπορέσουμε πράγματι να υιοθετήσουμε τις νέες ημερομηνίε εφαρμογής προκειμένου να μπορέσουμε να επιμείνουμε στους φιλόδοξους στόχους μας. Τώρα, πρωτού σας δώσω το λόγο κύριε Υπουργέ, θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό χρονικό σημείο εδώ, ε, σε ό,τι αφορά τον χάτη πορεία μας για την ολοκλήρωση της Οικονομικής ε, και Νομισματικής Ένωσης της ε, Ένωσης, καθώς αυτό αποτελεί βέβαια και μια ένδειξη της ισχύω του ευρώ, του κοινού μας νομίσματος και της ναι, μετά από μια περίοδο κρίσεων, σφαλμάτων και κακών αποφάσεων. Πολλοί δηλαδή λένε ότι τώρα η Οικονομική και Νομισματική Ένωση επανέρχεται στο προσκήνιο και από ό,τι γνωρίζω είσαστε μία από τις χώρες που επιθυμεί να προσχωρήσει στην Ευρωζώνη. Πράγμα βέβαια το οποίο είναι θετικό από την δική σας πλευρά και αποτελεί και μια ένδειξη ισχύω, αν θέλετε, του ευρώ και τη ευρωζώνη για μα. Οπότε θα ήθελα να σα ευχαριστήσω και για αυτή την πρόθεση από την πλευρά σα και για τα όσα θέλετε να κάνετε στο πλαίσιο τη ε, Βουλγαρική ε, Προεδρία. Αυτά από την πλευρά μου, αγαπητέ Βλάτισλαφ, σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας ε, σήμερα εδώ και θα ξεκινήσω με την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Προεδρίας μας στα βουλγαρικά. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη της ε, Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, η Βουλγαρία Βουλγαρία ήδη συμμετέχει στην ευρωπαϊκή οικογένεια κατά τελευταία 11 χρόνια και κατά τους επόμενους 6 μήνες θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί βέβαια το πολιτικό κέντρο του μηχανισμού λήψης αποφάσεων στην Ένωση. Ε, η δική μου αρμοδιότητα είναι τώρα να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας στον τομέα των οικονομικών υποθέσεων και η συνάντησή μας ε, σήμερα είναι σημαντική εν ώψη του οράματος που κατοχυρώνεται και στις συνθήκες ενός επικοδομητικού διαλόγου και της βελτίωσης της ε, θεσμικής συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως συνομοθετών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέρχεται μια ε, περίοδο σταθερή οικονομική ε, ανάπτυξη σε συνδυασμό με βελτιωμένε συνθήκε στην αγορά εργασία ε, και βελτιωμένε προποθέσει χρηματοδότηση. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα μία σειρά από προκλήσει και θεωρώ πω αν έχουμε μία υπεύθυνη στάση και αν έχουμε και ισορροπημένε πολιτικέ φιλοδοξίε, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει και να εξασφαλίσουμε μια γενικότερη οικονομική σταθερότητα και μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη καθώς και απασχόληση στην Ένωση. Εμείς ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω από την πλευρά της Βουλγαρικής Προεδρίας θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας σε ό,τι αφορά την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ε, εστιάζοντας σε μια σειρά από Την ολοκλήρωση της ε, Τραπεζικής Ένωσης, την περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών, την ε, περαιτέρω συζήτηση σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο για τους ε, δημοσιονομικούς κανόνες ε, και τις δυνατότητες σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μιας κοινή δημοσιονομικής ικανότητας αλλά και την ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ειδικότερα η Τραπεζική Ένωση αποτελεί μία από τις προτεραιότητε μας. Θέλουμε δηλαδή να εμβαθύνουμε το χάρτη πορείας που υπάρχει εδώ, προσθέτοντας κάποια συγκεκριμένα βήματα σε ό,τι αφορά τη μείωση του κινδύνου και την κατανομή του κινδύνου. Αυτό θα διευκολύνει και τη συζήτηση σε ό,τι αφορά ε, το κοινό backstop, ε, ε, αυτόν τον δημοσιονομικό μηχανισμό ασφαλείας, όπου βέβαια θα παίξει σημαντικό ρόλο και ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα. Ένα ακόμα ζήτημα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης. Ε, νομίζω πως το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει τις ε, εργασίες του σε ό,τι αφορά την ε, απλούστευση και την εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων, αλλά να ξεκινήσει και τις συζητήσεις για την εφαρμογή και τη μεταφορά στην νομοθεσία της Ένωσης, τη Σύμβασης, για τη, συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συνοσμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Με βάση την πρόοδο που θα επιτύχουμε σε αυτούς τους τομείς, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου ε, θα κληθεί να υιοθετήσει τον γενικότερο χάρτη πορείας για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ε, και θεωρούμε πως το πρόσφατο πακέτο της προτάσεων της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την ΟΝΕ αποτελεί μια πολύτιμη συνεισφορά. Κυρίε και κύριοι, η Βουλγαρική Προεδρία θα προσπαθήσει να επιτύχει την ομαλή εφαρμογή του κύκλου οικονομικού συντονισμού, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2018. Ε, το Συμβούλιο υιοθέτησε χθε ε, τα συμπεράσματά του σε ό,τι αφορά την ε, ετήσια έρευνα ανάπτυξης αλλά και την έκθεση μηχανισμού επαγρύπνησης και ενέκρινε τις συστάσεις σε ό,τι αφορά τον, την Ευρωζώνη. Ήθελα να σα ενημερώσω ότι θα ξεκινήσει ένα θεματικό διάλογο μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών το Μάρτιο του 2018 που θα εστιάσει ειδικότερα στι συστάσει του 2017 και όπου θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγικότητα τη εργασία. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την έγκριση από την πλευρά του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του πακέτου με τις συστάσεις αναχώρα για, για τα έτη 2018-2019 και βέβαια αυτό θα ενθαρρύνει την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αλλά και επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για το μέλλον τη Ευρώπη, εδώ ε, η ε, δημιουργία της Χρηματοοικονομικής Ένωσης ε, στο πλαίσιο ακριβώς της ολοκλήρωσης και της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης θεωρείται ως μία από τις βασικές προτεραιότητες και στην έκθεση των πέντε προεδριών αλλά και σε ένα από τα έγγραφα προβληματισμού της Επιτροπής σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης ε, που ε, ε, προτάθηκαν τον Μάιο του 2017. Όπως ήδη ανέφερα, μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης αλλά και της Προεδρίας μας είναι η περαιτέρω μείωση των κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα. Οι νομοθετικές προτάσεις που έγιναν από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2016 αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των μέτρων μείωση του κινδύνου. Η Εστονική Προεδρία έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο σε σχέση με τα τραπεζικά ζητήματα, αλλά παραμένουν μια σειρά από εκκρεμή ζητήματα πολιτική και τεχνική ε, φύση, για τα οποία θα χρειαστούν περαιτέρω προσπάθειε. Η Βουλγαρική Προεδρία έχει αναλάβει τη δέσμευση να ε, επιτύχει ένα ισορροπημένο συμβιβασμό σε σχέση με αυτά τα ζητήματα και ε, αναμένουμε να είμαστε σε να ξεκινήσουμε το διάλογο με το Κοινοβούλιο στο εγγύη μέλλον. Η πρόοδο που έχει επιτευχθεί. και θα πρέπει να επιτευχθεί είναι σημαντική καθώς ε, είναι προς το συμφέρον όλων των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρησιμοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες. Ε, θα εργαστούμε από εκεί και μετά ε, σκληρά προκειμένου να επιτύχουμε πρόοδο σε ό,τι αφορά την νομοθετική πρόταση, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων και βέβαια συμμορφούμενοι και με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το χάρτη πορεία για την ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ένωση ε, τον Ιούνιο του 2016, η συζήτηση σε ό,τι αφορά το πώ ακριβώ θα διαμορφωθεί αυτό το σύστημα ασφάλεια καταθέσεων θα ξεκινήσει μόλι θα έχουμε επιτύχει την επαρκή πρόοδο σε ό,τι αφορά τα μέτρα μείωση του κινδύνου. Ε, αυτή τη στιγμή μόνο τα κράτη-μέλη τη Ευρωζώνης ε, ε, συμμετέχουν σε όλα τα, τα στοιχεία, σε όλα τα επιμέρους τμήματα της Τραπεζικής Ένωσης, αλλά πάντοτε θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η πόρτα παραμένει ανοιχτή για όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, αλλά και ότι αυτό βέβαια συμβάλλει στη γενικότερη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα. Από εκεί και μετά, συνεχίζουμε τις εργασίες μας σε ό,τι αφορά την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών και θα συνεχίσουμε τις ε, συζητήσεις μας σε ό,τι αφορά νομοθετικές προτάσεις για τις υποχρεώσεις εκαθάρισης και την υποβολή εκθέσεων για τα παράγωγα, αλλά και σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενός ε, ε, πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξηγίαση των κεντρικών αντισυμβαλόμενων και τις ε, απαιτήσει ε, σε ό,τι αφορά τους σχετικούς ε, αντισυμβαλόμενους τρίτων χωρών. Ε, τώρα θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας σε ό,τι αφορά την πρόταση που έχει γίνει για ένα πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν προκειμένου να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή πρόοδο σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Η συζήτηση θα, η συζήτηση θα ξεκινήσει σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος ε, χρηματοοικονομικής εποπτείας ε, και σε ό,τι αφορά ένα νέο ε, καθεστώς ε, εποπτείας των επενδυτικών επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα την συμφωνία στην οποία φτάσαμε σε σχέση με τον κανονισμό για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών, τον ΕΜΗΡ δηλαδή. Είμαστε τώρα έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από την έγκριση βέβαια του Κοινοβουλίου της έκθεσής του με τις τροπολογίες που θα υποβάλει. Τώρα, ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα για τους ε, πολίτες μας είναι βέβαια, αλλά και τις επιχειρήσεις μας, είναι η φορολογία. Εδώ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στρατηγικά και ε, έγγραφα ε, χάρτη πορείας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά υπάρχουν και νομοθετικές προτάσεις που ήδη έχουν υποβληθεί και βέβαια θα λάβουμε υπόψη μας και τις γενικότερες πολιτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της Προεδρίας μας. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να προωθήσουμε τις επενδύσεις, να διασφαλίζουμε την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη αλλά και τον θέμητο ανταγωνισμό στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς μέσω ακριβώς δίκαιη και αποτελεσματικής φορολόγηση των εταιρικών κερδών που ε, προκύπτουν εντό τη Ένωση, ενώ θα προσπαθήσουμε βέβαια να καταπολεμήσουμε την ε, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και να αυξήσουμε την ε, φορολογική διαφάνεια. Μία ακόμα προτεραιότητά μας είναι βέβαια ο ευρωπαϊκός, ευρωπαϊκή ζώνη, αν θέλετε, ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος ΦΠΑ, ε, και εδώ θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στην χρήση αποτελεσματικών εργαλείων ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένη διαχείριση του ΦΠΑ προκειμένου να υπάρξει και καλύτερη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των αρμοδίων αρχών τους προκειμένου να καταπολεμηθεί η ε, απάτη σε σχέση με το ΦΠΑ. Ε, τώρα θα συνεχίσουμε και σε τεχνικό επίπεδο τις εργασίες μας σε ό,τι αφορά την κοινή ε, φορολογική ε, βάση εταιριών, ενώ και η φορολόγηση στις δομές της ε, ψηφιακής οικονομίας παραμένει σημαντική για μας. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μετά από την κατάρτιση της νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής, που την αναμένουμε δηλαδή αρχές του 2018, θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε πρόοδο το ταχύτερο δυνατό. Επίσης, στοχεύουμε στην διαμόρφωση μιας γενικότερης ε, προσέγγισης σε ό,τι αφορά την ε, οδηγία για τη διοικητική συνεργασία σε σχέση ειδικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ως προς ε, τις διασυνοριακές συμφωνίες. Και αυτό θέλουμε να το προωθήσουμε στο Συμβούλιο Κοφίν του Μαρτίου του 2018. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κοινή λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις μη συνεργαζόμενες ε, δικαιοδοσίες. Εδώ θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ε, και θα ε, προωθήσουμε δηλαδή τα αμυντικά μέτρα, τη διαδικασία διαγραφής από τη λίστα και όλα τα σχετικά πρότυπα. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσίασα τις κύριες προτεραιότητες της Προεδρίας μας και βέβαια το κλειδί για την επιτυχή εφαρμογή αυτών των προτεραιοτήτων βρίσκεται ακριβώς στην ενεργό και επικοδομητική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και είμαι πεπισμένο ε, ω προ τον σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, καθώ ε, προφανώς αποτελείται από τους εκπροσώπους των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια παίζει σημαντικότατο ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλή και πολύ σφαιρική η παρουσίαση που μας κάνατε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τα καλά σας λόγια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Μπάλτς είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω θερμά κύριε Υπουργέ εδώ στην ε, Επιτροπή ΕΚΟΝ. Χαίρομαι που βρίσκεστε σήμερα εδώ και θα ήθελα καταρχήν να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο για την Προεδρία σας, τόσο σε εσά προσωπικά όσο και στη χώρα σας για αυτό το πρώτο εξάμεινο του 2018. Δύο ερωτήματα θα ήθελα να σας θέσω. Το πρώτο είναι το εξής. Ως Προεδρία του Συμβουλίου, πώς ε, σκοπεύετε να διεξάγετε και να υποστηρίξετε τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο του Brexit, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το δικό μας τομέα των χρηματοοικονομικών ε, υπηρεσιών. Ποιε δηλαδή θα είναι οι προτεραιότητα σα ε, στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων. Δεύτερο ερώτημα. Ε, ο Πρωθυπουργό σα ε, πριν από μερικέ ημέρε προέβησε μια ανακοίνωση με βάση την οποία η δική σα χώρα προτίθεται να προσχωρήσει στην Ευρωζώνη. Τα δεδομένα τα οποία μα έχετε διαβιβάσει είναι εντυπωσιακά, αλλά υπάρχουν και κάποιε ανησυχίε, κάποιε σκέψεις δηλαδή ότι ενδεχομένως να υπάρχουν ακόμα κάποιες ελλείψεις. Ο Επίτροπος Μοσχοβησία ανέφερε για παράδειγμα ότι η παραγωγικότητα στη χώρα σας θα πρέπει να αυξηθεί αλλά και οι ξένε επενδύσει θα πρέπει να αυξηθούν. Άλλοι ανέφεραν ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα στο επίπεδο καταπολέμησης τη διαφθοράς. Οπότε εγώ θα ήθελα να σα ρωτήσω μπορείτε να μας δώσετε έτσι μια γενική επισκόπηση ως προς το ποια είναι τα μέτρα που, που θέλετε να λάβετε προκειμένου ακριβώς να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις. Ευχαριστώ. Να σας απαντήσω λοιπόν. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές και θα προσπαθήσω όσο μπορώ να απαντήσω και θα το κάνω με τη σειρά που κάνατε τις ερωτήσεις να σας πω πάντως πως ε, αισθάνομαι πιο άνετα μιλώντας για την κατάσταση στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή. Ε, καταλαβαίνετε ότι για μας η Ευρωζώνη και το Σέγγεν αποτελούν μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία για περαιτέρω ολοκλήρωση της ένταξης της Βουλγαρίας στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κάποιοι υποπτεύονται ε, πως ψάχνουμε εύκολα αποτελέσματα. Θέλω να σας καθησυχάσω. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν πως εμείς είμαστε μια χώρα που σέβεται τους δημοσιονομικούς κανόνες. Έχουμε τα μαθήματα που πήραμε από την μεταβατική εποχή, από το σοσιαλισμό, ε, στην σημερινή κατάσταση στη Βουλγαρία και αυτό μας, δί, μας δίδαξε ότι πρέπει με αυστηρό τρόπο να σεβόμαστε τους κανόνες. Έχουμε ε, το ΛΕΒ, το οποίο εδώ και 20 χρόνια είναι σε σταθερή οικονομία ε, με το ευρώ και για πρώτη φορά ε, το 1997 ξεκινήσαμε με σταθερές οτιμίες του ΛΕΒ με το Deutsche Mark είχαμε την πρώτη σταθερή οικονομία και μετά περάσαμε στη φάση που ε, αποκτήσαμε μια σταθερή οικονομία με το ευρώ. Και είναι κάτι το οποίο σεβόμαστε, επαναλαμβάνω εδώ και 20 χρόνια. Και έχουμε μάλιστα τη συναγματική οικονομία που είναι το 1,9553, σταθερότατο, και είναι το ίδιο το οποίο ίσχυε όταν περάσαμε από την ισοτιμία στο Deutsche Mark, στο Μάρκο Γερμανία, δηλαδή, ε, προ το ευρώ. Οπότε, να σας πω πως η δική μας κεντρική τράπεζα δεν έχει κανένα δικαίωμα έκδοσης διαφορετικό από αυτό το οποίο επιτρέπει στους υπόλοιπους η ΕΚΤ, οπότε θέλω να θεωρήσετε πως και εμείς είμαστε κομμάτι της αιμοδοσίας της Ευρωπαϊκής του ευρώ, γιατί μπορεί να είμαστε μεν ένα ξένο σώμα ως προς το ευρώ, αλλά και εμείς είμαστε υπό την πρέλα και τις πολιτικές επιλογές που κάνει η ΕΚΤ. Δεν είναι σαφές για μένα βέβαια τι θα έπρεπε να προπορεύεται Δηλαδή να πετύχουμε πρώτα την επαρκή σύγκληση και μετά να προσχωρήσουμε στην Ευρωζώνη ή αν η, ιδιότητα του μέλους της Ευρωζώνης θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι υπόλοιποι στην οικονομία μας και θα προωθήσει τις εξωτερικές επενδύσεις σε αυτήν. Και με τον τρόπο αυτό θα φτάσουμε στη σύγκληση. Μία από τις πιο πετυχημένες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η πολιτική συνοχής και η Βουλγαρία πρέπει να σας πω ότι όταν, προσχώρησε, όταν προσχωρήσει στην Ευρωζώνη θα προχωρήσει σε σύγκληση παρόλο που επαναλαμβάνω δεν βιαζόμαστε γιατί έχουμε ήδη τη στρατηγική στη θέση της και μιλάμε ήδη για τη συμμετοχή σε όλους τους μηχανισμούς ε, με πλήρη τρόπο αλλά επαναλαμβάνω η προσχώρηση στο ευρώ θα μπορούσε για μας κατ' επέκταση να θεωρηθεί πολιτική σύγκληση. Δεδομένου ότι εμείς δεν αποτελούμε κανένα κίνδυνο για την ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική. Το αντίθετο, θα ξέρατε κι εσείς πως η Βουλγαρία έχει το τρίτο χαμηλότερο ε, εξωτερικό χρέος και το πλεόνασμα το δικό μας είναι γύρω στο 1% του ΑΕΠ. Οπότε σε επίπεδο δημοσιονομικών κανόνων εγώ θεωρώ πως θα ήμασταν μάλλον μια θετική επιρροή και όχι μια αρνητική, ένα αρνητικό παράδειγμα για τους υπόλοιπους στην Ευρωζώνη. Φερνάντες. Όχι. Ο Άλφρεντ Σάντς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζουμε κύριε Υπουργέ. Καλή επιτυχία. Και να πω πως η πιο πρόσφατη αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης δείχνει πως η ανάπτυξη συνεχίζεται και στην Ευρωπαϊκή, ζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να μιλάμε πια για λιτότητα, δεν χρειάζεται πια να ζητάμε περικοπές ε, από τη μεσαία τάξη και από ε, τους συνταξιούχους, άρα μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυξήσεις μισθών. Να έχουμε μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και να μειωθούν οι ανισότητες. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυξήσει της τάξης του 5% στους ελάχιστους ε, μισθούς όπου αυτοί ισχύουν. Έτσι ώστε και οι ανταγωνιστικές πιέσεις να εξισορροπηθούν και να πετύχουμε όλοι τους στόχους μας με τα νομισματικά εργαλεία διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιεί η τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό πρέπει να το αποφασίσει το Συμβούλιο. Πιστεύετε πως υπάρχει κάποιος που να έχει όρεξη να κάνει κάτι τέτοιο γιατί ξέρετε πως σύντομα θα γίνουν βουλευτικές εκλογές στα κράτη-μέλη ε, και επειδή θα γίνουν και ε, ε, εκλογές για τους ευρωβουλευτές πιστεύω πως θα πρέπει να αποδείξουμε ότι θέλουμε να ζουν καλύτερα οικογένειες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάτι διαφορετικό. Αφού λύγει η, Ευρωπαϊκή, η θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πείτε μου, τι πιστεύετε του Εύση και η πολιτική συνεχή ήταν πετυχημένα φέραν σύγκληση μεταξύ των οικονομιών του κέντρου και της Ανατολής και της περιφέρειας γενικότερα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές ερωτήσεις σαν αυτές που μου κάνετε και πιστεύω πως θα μπορούσαμε να μιλάμε για τα θέματα αυτά για μέρες. Λιτότητα και μέτρα λιτότητας. Να ξεκινήσουμε εκεί. Νομίζω πως οι τρέχοντες δημοσιονομικοί κανόνες είναι εξαιρετικά περίπλοκοι και θα πρέπει να συζητηθούν σε επίπεδο συμβουλίου και θα πρέπει να απλουστευτούν, αυτό είναι το βέβαιο για τις δημόσιες δαπάνες μπορεί να προκαλέσουν προστιθέμενη αξία, αλλά έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα με τις οποίες θα τις χειριστούμε. Και πρέπει να παραδεχτούμε το εξής, όπου οι δημόσιες δαπάνες ε, για τη στήριξη εισοδημάτων ε, έχουν εφαρμοστεί, αυτό έχει γίνει με διόγκους του εθνικού προϋπολογισμού και εις βάρος της ανταγωνιστικότητας, γιατί ξέρετε πως το μέσο χρέος στην Ευρώπη είναι αρκετά υψηλό. Και αν αυτή τη στιγμή ε, προχωρήσουμε σε αύξηση των δαπανών εις βάρος των επόμενων γενναιών, θα καταλήξουμε σε κάτι το οποίο είναι άδικο. το να αυξήσουμε τις δαπάνες και να συνάψουμε περισσότερα δάνεια δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση για την βουλγαρική κυβέρνηση. Για την ανάπτυξη, ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε σε μια φάση ανάπτυξης και στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη πιστεύουμε ότι αυτά μπορούν να φέρουν πολλά θετικά. Αυτή τη στιγμή όμως δυστυχώς επειδή ε, βρισκόμαστε στη φάση της ανάκαμψης θα πρέπει τώρα να προλάβουμε την ενδεχόμενη ε, επόμενη στροφή του κύκλου και να προλάβουμε ε, μια αρνητική φάση και θα πρέπει ως φρονίμων τα παιδιά να κάνουμε κάποιες προσπάθειες έτσι στην επόμενη κυκλική φάση της οικονομίας να είμαστε πιο έτοιμοι. Τώρα, να σας δώσω κάποια ε, παραδείγματι, Βουλγαρία πριν από 10 χρόνια ε, το μέσο ΑΕΠ ε, στη Βουλγαρία ήταν στο 26% και λόγω της πολιτικής σύγκλησης και της αλληλεγγύης και της ιδιότητας του μέλους φτάσαμε να έχουμε ένα μέσο ΑΕΠ και σας δίνω στοιχεία του 16 40% των υπολείπων κρατών μελών. Οπότε περάσαμε από το 1 τρίτο σε περίπου το 1 δεύτερο του μέσου ΑΕΠ της Ευρώπης. Οπότε αυτό αποτελεί πολύ σημαντική πρόοδο και για τους δικούς μας πολίτες η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μεγάλη επιτυχία. Και είμαι σίγουρος πως ο ρόλος τον οποίο έχουν παίξει οι Εθνικοί Υπουργοί Οικονομίας σε σχέση με τα θέματα αυτά έχει να κάνει με τις εθνικές παραδόσεις, με τις κομματικές ε, θέσεις, αλλά δεν πιστεύω πως η αύξηση ε, προϋπολογισμών ε, ε, θα είναι μια λύση η οποία μπορεί να ισχύσει στο ειδηνικές. Thank you. Ευχαριστώ. Kate Winburn. Καλημέρα, καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ και σας ευχαριστώ που ήρθατε να μας μιλήσετε σήμερα. Η ερώτησή μου αφορά τη συνέπεια των κανόνων που έχουμε στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή και το Συμβούλιο σας διαπραγματεύτηκαν τρεις ε, φακελούς όσον αφορά τα παράγωγα και τι υπηρεσίε εκαθάριση. Και όπω είπατε υπάρχει το σύστημα επίλυσης διαφορών και τον κανονισμό ε, του REFIT και τον εποπτικό μηχανισμό. Ως ε, εισηγήτρια του πρώτου θέματος που σας ανέφερα γνωρίζω ότι υπάρχουν προκλήσεις και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται στον πρώτο κανονισμό δεν ε, είναι εις βάρος των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν από άλλο κανονισμό και ορισμένες φορές έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα τι κάνετε για να υπάρχει συνέπεια στα τρία θέματα αυτά. Και δεύτερον, αυτό είναι αρκετά δύσκολο ούτω ή άλλω, αλλά εάν προσθέσουμε και το Brexit, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ σύνθετα. Πώ θα διασφαλίσει λοιπόν ότι η Βουλγαρική Προεδρία ότι οποιαδήποτε δράση λάβουμε και κυρίω ό,τι αποφάσει λάβουμε για τα θέματα αυτά δεν θα υποσκάψουν και δεν θα. Ε, προδικάσουν αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν όσον αφορά το Brexit. Ιδίω όταν αφορά το θέμα της ε, ε, ε, φορολογικές βάσεις τρίτων χωρών και πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα υπάρχει συνέπεια με τα όσα συζητούνται με τις διαπραγματεύσεις με το Brexit στην Task Force. Ευχαριστώ. това е една Το Brexit είναι λυπηρό γεγονός και λυπάμαι που οι Βρετανοί πολίτες ψήφισαν με τον τρόπο που ψήφισαν, διότι είμαι βέβαιος ότι εντός της Ένωσης ε, διασφαλίζεται η ειρήνη στην Ήπειρο και δεύτερον, οι διαιρέσεις στην παρούσα οικονομία δεν αποτελούν καλή ιδέα. Οι μικρότεροι θα γίνουν πιο αδύναμοι και οι πιο ισχυροί θα γίνουν ακόμα πιο ισχυροί. Όσον αφορά τα θέματα που αναφέρετε, θεωρούμε ότι είναι νέο ε, πακέτο. Οι εμπειρογνώμονε μας ασχολούνται ταυτόχρονα με τα θέματα αυτά για την πρόταση για την εποπτεία και τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους και το θέμα για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους εξετάζεται και ως τμήμα του κανονισμού για τις ε, ε, υποδομές της αγοράς. Αυτά όλα συζητώνται ταυτόχρονα στις ομάδες εργασίας στο Συμβούλιο. Ε, βάσει και των όσων έχουν επιτύχει οι Εστονοί, Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε σημαντική πρόοδο για την πρόταση για την εποπτεία του κεντρικού αντισυμβαλόμενου και ε, η αναθεώρηση του σχεδίου για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους ε, στην, ε, στον κανονισμό για τις υποδομές των αγορών νομίζω ότι θα ενταχθεί καταλήλων. Εγώ είμαι με τριοπαθώ αισιόδοξο και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε όλα αυτά όσον αφορά του ε, τους τρίτους. Τον Οκτώβριο, στη διάρκεια της Εστονικής Προεδρίας, ε, καταλήξαμε σε συμφωνία για την ε, διαπραγματευτική εντολή για το ΕΜΙΡ και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε συζητήσεις μόλις είναι έτοιμο και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλίντς. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προχωρήσει αρκετά σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες, για παράδειγμα σε σύγκριση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Αναφέρομαι εδώ ιδιαίτερα στο διαδίκτυο και σε άλλες τέτοιες τεχνολογίες και αν πραγματικά θέλουμε να είμαστε ένας από τους ηγετικούς οικονομικούς χώρους στον κόσμο, τότε θα πρέπει ακριβώς να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος, ε, όχι μόνο σε, αυτές, σε σχέση με αυτές τις τεχνολογίες, αλλά και σε ό,τι αφορά την κινητικότητα. Αλλά εγώ δεν άκουσα τίποτα στη δική σας παρουσίαση σε σχέση με αυτό το ζήτημα, οπότε ε, θα υπάρξουν προτάσεις στο πλαίσιο της δικής σας ε, προκειμένου να επιτύχουμε περισσότερες επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς και έτσι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το γεγονός ότι λόγω της αποχώρησης με τον Brexit του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε λιγότερα κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρότι όμως αυξάνονται οι δαπάνες της. Όχι μόνο ε, των δαπανών σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ε, ανάπτυξη αλλά και σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό ζήτημα και τις διαφορετικές δαπάνες που έχουν προκύψει σε αυτό το πλαίσιο. Άρα λοιπόν μήπως θα έπρεπε τώρα να προβείτε σε μια επανεξέταση της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών μελών και ένωσης. Δηλαδή αναφέρομαι ειδικότερα στην αρχή της επικουρικότητας ε, δηλαδή ουσιαστικά να αντλήσουμε τα διδάγματα που θα έπρεπε έτσι ώστε να πούμε ότι κατανέουμε τέτοιο τρόπο τις αρμοδιότητές μας ε, προκειμένου τα κονδύλια να επαρκούν για τις προτεραιότητές μας. Ένα ακόμα ζήτημα. Ε, γνωρίζουμε πως πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάστηκε να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και να επανακατασταθούν στη Βουλγαρία και για φορολογικούς βέβαια λόγους. Αυτή η διαδικασία έχει σταματήσει τώρα, έχει διακοπεί ή συνεχίζεται ακόμα. καθώς ε, αφού και η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε φάση ανάκαμψης ε, δεν θα έπρεπε να σταματήσει αυτή η διαδικασία αφού αποτελεί βέβαια και ε, πρόβλημα σε δημοσιονομικό επίπεδο για την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Πράγματι το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ δεν μπορεί να θέσει ως προτεραιότητα το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορώ να σας πω το εξής όμως. Θυμάμαι ακόμα την επιτυχή ε, απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να συνεργαστεί με τη γαλλική κυβέρνηση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να ξεκινήσει το πρόγραμμα Άβης συγγνώμη. Ε, πρόκειται για ένα project που ουσιαστικά αμφισβήτησε την υπεροχή των ε, ε, κυρίαρχων Αμερικανικών εταιριών. πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή των ε, ε, τεχνολογιών. Η Ευρώπη πριν από 10 χρόνια ε, βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας. Θυμόμαστε όλες τις εφευρέσεις οι οποίες ξεκίνησαν από τη γυραιά Ήπειρο. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Στις μέρες μας ε, είναι άλλοι ε, στην πρώτη γραμμή, αλλά για μας ε, στο Συμβούλιο Κοφίν η προτεραιότητά μας είναι η φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας και το θέμα της φορολογίας είναι πρώτη προτεραιότητα για μας πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να φορολογήσουμε τις πολυεθνικές επιχειρήσεις μέσω φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας ε, θα μπορέσουμε ίσως να εξεύρουμε και τρόπους να φορολογήσουμε πολυεθνικές επιχειρήσεις ώστε τα κέρδη τα οποία ε, δημιουργούνται στην Ευρώπη θα παραμένουν στην Ευρώπη προς όφελος των πολιτών μας. Ε, το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι πιο διάφανο και πιο δίκαιο. Τώρα, Έχουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου του 2017 και είμαστε και εν αναμονή των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΣΑ, της έκθεσης του ΟΣΑ. Ε, κατά πάσα πιθανότητα θα τα λάβουμε τον Μάρτιο του 2018 και θα ξεκινήσει η αξιολόγηση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αμέσως ε, μετά την παραλαβή τους. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις και το ενδεχόμενο μηδενικής φορολόγησής τους. Πρόκειται για μία πρόταση που ακόμα είναι υποσυζήτηση. υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ δύο κρατών μελών και αυτό οδήγησε σε μπλόκο της συγκεκριμένης συζήτησης το 2017. Όσον αφορά τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων από την Ελλάδα στην ε, Βουλγαρία, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει ε, κάποια α, ως αντίκτυπος ε, στη Βουλγαρία, δεν ήταν τόσο μεγάλη αυτή η μετεγκατάσταση. Και βεβαίως εμάς ο στόχος μας είναι να υπάρχει ένα δίκαιο σύστημα φορολόγησης και όσον αφορά τους ε, φορολογικούς συντελεστές και όσον αφορά τη φορολογική βάση. Ε, είναι πολύ ε, ευπρόσδεκτη η ανάκαμψη της Ελλάδος και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Θεωρούμε ότι ο αντίκτυπος δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήσαμε γέρος, αλλά πρέπει να σεβόμαστε και το χρόνο των 5 λεπτών για κάθε ερώτηση και απάντηση, Αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όλου. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από τα μέλη να μιλούν για 2 λεπτά το πολύ και 3 λεπτά για τον ε, καλεσμένο μα ε, για να απαντήσει. Ο κ. Παπαδημούλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. σα καλωσορίζω κύριε Υπουργέ και εύχομαι καλή επιτυχία στη Βουλγαρική Προεδρία. Σας ευχαριστώ και για τα θετικά σχόλια που μόλις κάνατε για την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας μου της Ελλάδας, θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής. Από ό,τι είδα ήδη χθες στο ΕΚΟΦΗΝ, θέσατε ως μία από τις προτεραιότητες την, ε, τον κοινωνικό πυλώνα. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις ήδη και κάποιες αποφάσεις στο Γκότεμπουργκ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και με ποιο χρονοδιάγραμμα σκοπεύετε να πάρετε για την ε, ενίσχυση του κοινωνικού πυλώνα. Το δεύτερο, με ικανοποίηση άκουσα ότι είναι ψηλά στις προτεραιότητές σας η προώθηση της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και μάλιστα με μια παράλληλη προσέγγιση, μείωση κινδύνου, κατανομή κινδύνου, παράλληλα έτσι ώστε να διαμορφωθεί αυτό το κοινό backstop. Εν ώψη του ECOFIN του Μαρτίου θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να προχωρήσει αυτό το θέμα, δεδομένου ότι το θέμα αυτό υπάρχει μια μακρόχρονη καθυστέρηση με ευθύνη του Συμβουλίου. Το τρίτο θέμα αφορά στον πολιετή προϋπολογισμό της Ένωσης ε, εν ώψη και του Brexit πώς αξιολογείται την πρόταση να υπάρξουν και νέοι πόροι στον κοινοτικό προϋπολογισμό με δεδομένο ότι υπάρχουν σαφείς κίνδυνοι για δραματικές περικοπές επικίνδυνες για την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή στα κονδύλια και της συνοχής και της κοινή αγροτικής πολιτικής. Ποια είναι η προσέγγιση της Προεδρίας της Βουλγαρίας στο θέμα αυτό. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολιετής ε, δημοσιονομικές προοπτικές να σας πω πως εδώ <laughs> είναι μάλλον οδυνηρή η συζήτηση που έχουμε να κάνουμε στα πλαίσια του Brexit και η συζήτηση και οι συζητήσεις μάλλον δεν έχουν εστιάσει τα σωστά σημεία. Χρειαζόμαστε να ξέρουμε ποιες είναι οι πολιτικές που θα χρειαστούμε, ποια είναι τα μέσα και τα εργαλεία και μετά να τους δώσουμε σάρκα και οστά. Είναι πολύ διαφορετικές οι απόψεις και να σας πω πως το Μάρτιο στη Σόφια θα κάνουμε μια συζήτηση υψηλού επίπεδου ακριβώς για το θέμα των πολιετών αυτών προοπτικών. Δεν νομίζω πως τα κράτη-μέλη επιθυμούν να δημιουργήσουμε νέα μέσα για να καλύψουμε αυτό το μελλοντικό κενό και με σκεπτικισμό αντιμετωπίζω ε, τη δυνατότητα με τα τρέχοντα μέσα να είμαστε σε θέση να αυξήσουμε τις συνεισφορές των καθαρών εισφορέων Και τώρα για όσους λαμβάνουν ε, κονδύλια και από την ΚΑΠ και από τα Ταμεία Συνοχής, νομίζω πως τα δύο αυτά μέσα είναι πολύ σημαντικά, πολύ ευνοϊκά, είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικά, έχουν δείξει τι αξίζουν και η συζήτηση θα είναι δύσκολη. Και βέβαια περιμένουμε χαρά προτάσεις από την Κομισιόν για τα θέματα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει το σημαντικό είναι να εγκριθούν από εσάς στην τρέχουσα θητεία από την Επιτροπή σας γιατί αν το αναβάλουμε υπερβολικά μετά τις ευρωεκλογές δηλαδή οι συζητήσεις θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολες νέοι επίτροποι, νέοι ευρωβουλευτές και θα ξεκινήσουν και πάλι από μηδενική βάση όλες αυτές οι συζητήσεις. Για το θέμα τώρα της ενίσχυσης της Οικονομικής και της Νομισματικής Ένωσης στηρίζουμε απόλυτα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα και ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η συζήτηση που έγινε. Να σας πω πως το πακέτο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ χρήσιμο. Πιστεύω πως αποτελεί μια πολύ θετική συμβολή τουλάχιστον μακροπρόθεσμα. Και το Συμβούλιο συζήτησε το θέμα μετά τις συζητήσεις εκεί είπαμε θα παραμείνουμε σε επαφή με τον Μάριο Σεντένο που είναι πρόεδρος πλέον της Ευρωζώνης έτσι ώστε να επιτύχουμε το υψηλότερο επίπεδο συντονισμού γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά τα αμφιλεγόμενα θέματα και εδώ πρέπει να δούμε τι θα γίνει και ποια προτεραιότητα θα τηθεί risk sharing ή risk reduction δηλαδή μείωση κινδύνου ή αμοιβαιοποίηση αυτού Κάποιοι θέλουν να προχωρήσουμε βήμα-βήμα, πρώτα μείωση κινδύνου και μετά, αφού σημειώσουμε πρόοδο, να περάσουμε στην κατανομή αμοιβιοποίηση του κινδύνου και να σας πω πως αυτό είναι ένα εξαιρετικά ακανθώδες θέμα για το οποίο όμως κρατημέλη θέλουν να σημειώσουμε πρόοδο. Ο κύριος Ούρτανσον. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που, έρχεται, που ήρθατε σήμερα. Έχω πολύ συγκεκριμένα και σύντομα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, η ομάδα μου ανησυχεί γιατί τους τελευταίους μέσες ε, έχουμε πολλά προσκόμματα για την Τραπεζική Ένωση και για τα όσα γίνονται για τις διασώσεις τραπεζών. Για το πακέτο αυτό, το Risk Reduction, πείτε μου τι γίνεται και πείτε μου αν αυτά τα εμπόδια που διαπιστώσαμε να υπάρχουν ε, πρόσφατα ε, έχετε κάποια πρόταση για να ξεπεραστούν. Αυτό. Δεύτερο. Στα έγγραφα που υπέβαλε η Προεδρία και δεν τον αναφέρατε ούτε εσείς καμία αναφορά στην πρόταση της ε, αναθεώρηση οδηγία για την ανακράτος μέλος ε, έκθεση. Τι θα γίνει, μέσα στο εξάμεινο θα το δείτε, έχετε την πρόθεση να το βάλετε στα σκαριά. Και η τρίτη ερώτηση σχετίζεται με κάτι που είπατε, ο, το περίφημο μαύρο κατάστοιχο με τους ε, φορολογικούς παραδείσους. Εμείς, πολλοί είμαστε εμείς που δεν συμφωνούμε με τα όσα αποφάσισε χθε ο ΕΚΟΦΗΝ. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Γιατί δεν έχουμε κανένα ε, επιχείρημα. Για ποιο λόγο βγάλαν κάποιος από τον κατάλογο αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε. Εσείς είστε η Προεδρία. Τι πιστεύετε. Τα έγγραφα τα οποία, στα οποία βασίστηκε η απόφαση να βγάλουμε κάποιες χώρες θα πρέπει να είναι δημόσια. Τουλάχιστον να έχει πρόσβαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί μια τέτοιου είδους απόφαση χωρίς να δικαιολογείται και να τεκμηρώνεται τουλάχιστον ε, σε εμά εδώ, ε, προκαλεί ανησυχία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια ως προς την διαδικασία συμπερίληψης ή διαγραφής από τη λίστα μιας χώρας. Και αυτό βέβαια και για λόγους συνεργασιμότητας από την πλευρά αυτών των χωρών. Η εν λόγω δηλαδή η διαδικασία θα πρέπει να είναι παρκώς δημόσια έτσι ώστε να είναι και παρκώς αξιόπιστη. Θα αναφέρει ότι δεν θα ήταν κακό το να δημοσιεύσουμε τις ε, χώρες ε, οι οποίες διαγράφηκαν από τη λίστα. Ωστόσο, ε, με βάση το, τα όσα προβλέπει η διαδικασία, θα πρέπει οι εν λόγω χώρες να ε, δώσουν τη συνένεσή τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκύψει ένα διπλωματικό πρόβλημα ανάμεσα στα αυτά τα κράτη-μέλη δηλαδή και τις μη συνεργαζόμενες χώρες. Μπορώ ωστόσο να σας διαβεβαιώσω ότι η ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου του Συμβουλίου εξετάζει πάρα πολύ προσεκτικά τις ε, δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι χώρες οι οποίες διαγράφηκαν από τη λίστα και βέβαια επιφυλασσόμαστε να επαναφέρουμε στη λίστα αυτές τις χώρες εφόσον δεν ανταποκριθούν σε αυτές τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβαν. Δηλαδή ουσιαστικά να τις ε, θεωρήσουμε και πάλι ως μη συνεργαζόμενες ε, περιοχές δικαιοδοσίας. Νομίζω πως ε, αυτό καταδεικνύει πως η απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο είναι θετική. Οι χώρες δηλαδή οι οποίες συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν τον κατάλογο πολύ γρήγορα ανέλαβαν τι σχετικέ ε, δεσμεύσει, αποφάσισαν δηλαδή να συνεργαστούν μαζί μα. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι πράγματι ήταν σωστή απόφαση που λάβαμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, υποβολή εκθέσεων, σε ό,τι αφορά τι ε, τρίτε χώρε, οι σχετικέ εργασίε προωθήθηκαν αρκετά στο πλαίσιο της Ολλανδικής, της Εθνική ε, Προεδρία ε, και άλλων, τη ε, και νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε πιο σαφής τώρα ως προς τις διατυπώσει μα εδώ γιατί και η νομική υπηρεσία αναφέρει πως η νομική βάση θα πρέπει να είναι το άρθρο 15 ενώ η άλλη άποψη είναι από νομική βάση θα πρέπει να είναι το άρθρο 50α της συνθήκης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει συνάντηση σε επίπεδο Συμβουλίου ως προς αυτό. Ευχαριστώ κύριε Σκόμπορν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το 2007 η ε, Βουλγαρία ήθελε να προσχωρήσει στην Ευρωζώνη αλλά δεν πληρούσε τα σχετικά ε, κριτήρια αλλά βέβαια γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να αποφασίσετε το τι επιθυμείτε από αυτά τα προνόμια. Δηλαδή θα πρέπει να πληρείτε όλες αυτές τις προϋποθέσεις ε, σε ό,τι αφορά τη, ε, τη σταθερότητα και ό,τι καθεξής. Και ουσιαστικά θα υπάρχει ένας Υπουργό Οικονομικών της Ένωσης ο οποίος θα είναι αρμόδιος για τα δημόσια οικονομικά σας και όχι εσείς ε, πλέον. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θα καταστραφεί η ανταγωνιστικότητά σας, δεν θα μπορείτε να είστε ανταγωνιστικοί ως χώρα και έχετε φορολογικό συντελεστή τάξη του 10% επί των εταιρεών. Ουσιαστικά είναι ε, μια πάρα πολύ όμορφη κατάσταση όπως ισχύει στη χώρα σας αυτή τη στιγμή. Ε, γιατί α, θέλετε τώρα να το αλλάξετε. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι θέλει τώρα αυτή η ενωπημένη βάση φορολόγηση των εταιρεών συνδυαστεί με έναν κοινό φορολογικό συντελεστή για όλους. Ουσιαστικά είναι κάποιοι οι οποίοι, οι γραφειοκράτες οι οποίοι θα λάβουν αυτές τις αποφάσεις και θα υποφεληθούν από αυτό, όχι οι πολίτες. Και εάν υπάρξουν ε, πράγματι κάποια, κάποια διακριτική μεταχείριση όπως αυτή ε, προβλέπεται για, την, ε, για το Λονδίνο, τότε ενδεχομένως να υπάρξουν προβλήματα και για κάποιες αμφιβόλου αξιοπιστίας ιταλικές τράπεζες που σημαίνει με τη σειρά του αυτό ότι θα υπάρξουν και για την Ευρωζώνη. Εμείς δεν σημαίνει επειδή αποχωρούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω θέλουμε να βιώσουμε μια καταστροφή της Ευρωπαϊκής Ένωση, όπως αυτή που είχαμε δει το 1929 και άλλο τέλα. Ουσιαστικά με τον τρόπο ε, που τα πράγματα συμβαίνουν και με την προσχώρηση τη τώρα στην Ευρωζώνη ουσιαστικά ε, κινείστε προ αυτή την κατεύθυνση. επειδή έχω συμμετάσχει και στα, όσα διαχειρίζεται το Λονδίνο σε αυτό το επίπεδο, ε, γνωρίζω ε, γιατί μιλάω. η, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση υπονομεύει ουσιαστικά μία σειρά από χώρες, για παράδειγμα, μέσω και της, ε, ε, τα όσα έχει κάνει σε σχέση με την εισβολή στην Ουκρανία και αλλού. Τον διακόπτη τον ομιλητή ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας με την οποία ωστόσο δεν ε, συμφωνώ. Εγώ υποστηρίζω πλήρως την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ πως ε, ε, το Brexit είναι μια δυσάρεστη υπόθεση. Αλλά προφανώς αυτή ήταν η βούληση του εκλογικού σώματος της Μεγάλης Βρετανίας. Γνωρίζετε πως η δική μου θέση είναι ότι η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας σημαίνει πως ε, οι ισχυροί παίκτες θα καταστούν ακόμα ισχυρότερα. Ενώ οι πιο αδύναμοι θα χάσουν ακόμα περισσότερο σε δύναμη. Θα δούμε βέβαια, η ιστορία θα δείξει κατά πόσο έχουμε δίκιο ή όχι, αλλά ε, η επιβολή μιας ενοποιημένης κοινής φορολογικής βάσης για τις εταιρείες δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα αρμονισμένος φορολογικός συντελεστής. Μπορούμε να έχουμε με ενοποιημένη κοινή βάση ανεξαρτήτω και ελπίζουμε ότι πραγματικά θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και να επιτύχουμε πρώτα. Με αυτόν τον ε, τρόπο θεωρούμε πως ε, θα υπάρξει πιο δίκαιη μεταχείριση των επιχειρήσεων χωρίς να υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τον ε, φορολογικό ανταγωνισμό. Δεν θέλουμε δηλαδή ε, δεν, δεν θεωρούμε πως θα υπάρξει πρόβλημα σε ό,τι αφορά και τη δική μας ε, ε, προσχώρηση στην Ευρωζώνη. Δεν βλέπω, δηλαδή, δεν αντιλαμβάνομαι τις αντιστοιχίες που μας εκφράσατε. Έχουμε μια πολύ, ε, ένα πολύ καλό οικονομικό επιτελείο το οποίο εξέτασε αυτά τα ζητήματα και δεν θεωρούμε ότι προκύπτει ένας κίνδυνος δημοσιονομικού χαρακτήρα για τη Βουλγαρία. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι πού βασίζεται τη δική σας τοποθέτηση και σε καμία περίπτωση τις μέσες που θα αναλάβουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο ε, στην ε, Ένωση. Κύριε Κάπελ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην ε, Προεδρία σας και βέβαια αυτό το λέω και για δικό μου όφελος γιατί είμαι προφανώς επίκοσης της Αυστρίας οπότε η επόμενη Προεδρία του Συμβουλίου είναι η δική μας και αν η δική σας προεδρία στεφτεί με επιτυχία, τόσο το καλύτερο βέβαια και για τη δική μας. Τώρα, μας παρουσιάσατε σήμερα εδώ ορισμένε από τις προτεραιότητες της προεδρίας σας, ε, μεταξύ αυτών η καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής, ε, μέτρα για την περισσότερη διαφάνεια και την καλύτερη διοικητική συνεργασία ειδικότερα στον χώρο του ΦΠΑ αλλά υπάρχουν από εκεί και μετά και μια σειρά από ζητήματα εναρμόνισης σε ό,τι αφορά την κοινή βασιολόγηση εταιρεών και την ενοποιημένη κοινή βασιολόγηση εταιρεών. Εμείς όπως γνωρίζετε ε, πως ε, είμαστε και εμείς όπως εσείς σε μια χώρα σχετικά ανοιχτή σε ό,τι αφορά τους ευρωλογικούς συντελεστές οπότε θα ήθελα να μας πείτε ε, πώς θα μπορέσετε με τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία να επιτύχετε πρώτο σε σχέση με αυτές τις προτεραιότητες. Δεύτερο ζήτημα ε, η υποψηφιότητά σας ε, για την ε, προσχώρηση δηλαδή στην Ευρωζώνη, γιατί μόλι τώρα μα είπατε ότι θα υποβληθεί επίσημα και ένα αίτημα συμμετοχής μέσα σε αυτό το εξάμεινο. Πράγματι, συνοδεύεται και από καλά δημοσιονομικά στοιχεία, έχετε δηλαδή δημοσιονομικό πλεόνασμα, ε, έχετε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, ε, γύρω στο 4%, αλλά ταυτόχρονα το κατακεφαλή ΑΕΠ ε, βρίσκεται κατά 18% χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε να συγκεντρώσετε την απαραίτητη πλειοψηφία στο επίπεδο του Συμβουλίου ούτως ώστε δηλαδή να υπερψηφίσουν αυτή την προσχώρηση, ειδικότερα σε ό,τι αφορά ε, και την καλύτερη ποιότητα ζωής και την εξασφάλιση ίσων όρων παιχνιδιού για όλους. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την Προεδρία, σας διαβεβαιώ ότι θα σας αφήσουμε και εσάς δουλειά, μην ανησυχείτε. Είμαστε σε επαφή με τον Υπουργό Οικονομικών σας. Ε, είναι πάρα πολύ επικοδομητικός ο διάλογος. Το Φεβρουάριο στη Βιέννη θα υπάρξει και μια συνάντηση των τριών Υπουργών ε, του Τρίου, της Εστονίας, ε, της Αυστρίας και του δικού μας. Και όλοι θα δούμε τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Προκλήσεις που είναι κοινές όσον αφορά τη βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης ε, που εξαρτάται φυσικά από την ποιότητα της διακυβέρνησης και εμεί ω κυβέρνηση ε, κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες ε, προκειμένου να βελτιώσουμε το βουλγαρικό βιωτικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια η αύξηση του εισοδήματος ήταν διψήφια και αυτό μας οδηγεί κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο εισοδήματος και ελπίζουμε να προχωρήσει πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία. και φαίνεται να υπάρχει και μείωση της μετανάστασης ε, των ε, Βουλγαρών. Είναι μικρότερη από ό,τι στο παρελθόν. Για μας λοιπόν θα θεωρηθεί ιδιαίτερη επιτυχία να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα κατάλληλο βιωτικό επίπεδο που θα προσελκύει μετανάστες και όχι το αντίστροφο υπάρχουν και αρκετοί ηλικιωμένοι Ευρωπαίοι οι οποίοι έχουν ε, ε, μετακομίσει στην ε, Βουλγαρία μετά τη συνταξιοδότησή τους. Έχουμε οικογένειες από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα και από την Αυστρία. φαίνεται λοιπόν να είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν τη σύνταξή τους στην Βουλγαρία. Έχει πολύ ωραία φύση η Βουλγαρία και σίγουρα το κλίμα είναι πολύ καλύτερο από τις Βρυξέλλες. Thank you, Darius Rosati. Ευχαριστώ, Ντάριο Ροζάτη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλωσορίσατε στη συνεδρία της Επιτροπής ΕΚΟΝ και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία ε, ως Πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι για τις απώλειες ε, που ε, αντιμετωπίζουν ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη φορο... αποφυγή ΦΠΑ. Χάνονται εκατομμύρια κάθε χρόνο λόγω παραπλανητικών συναλλαγών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ε, ψευδών συναλλαγών. Ε, έχουμε και μία έκθεση μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το οριστικό ε, φορολογικό σύστημα ΦΠΑ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ασχοληθεί με αυτές τις απώλειες που μόλις σας ανέφερα και σε τι βαθμό θα μπορέσουμε να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής για κακές πρακτικές ΦΠΑ. σκοπεύετε να αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες ε, ώστε να μπορέσετε να καταπολεμήσετε αυτές τις ε, πρακτικές, ε, πρακτικές οι οποίες στοιχίζουν τόσα πολλά για τα κράτη-μέλη μας. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τα αποτελέσματα της εργασίας της ειδική Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Κοινοβουλίου για τα Panama Papers. πρόκειται για μια ad hoc επιτροπή η οποία παρουσίασε τα αποτελέσματά της στο Κοινοβούλιο. Η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ενέκρινε τις συστάσεις ε, και θέλουν να μειώσουν το πεδίο φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής και ξεπλήματο. Ε, τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν εσείς ώστε να εφαρμοστούν αυτές οι συστάσεις. Είστε διατεθειμένος ε, να προχωρήσετε το θέμα αυτό. Някои изследвания показват, че годишно загубата Υπάρχουν έρευνες οι οποίες καταδεικνύουν ότι οι αιτήσει απώλειες ΦΠΑ ισοδυναμώνουν με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. 150 δις το 2015. Η Βουλγαρία με την Αυστρία, την Τσεχία και την Ουγγαρία ξεκίνησαν μία πρωτοβουλία προκειμένου να τροποποιηθεί η οδηγία ΦΠΑ θέλαμε να ε, συμπεριληφθεί ο μηχανισμός αντίστροφης ε, χρέωσης ε, για πολλά προϊόντα. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υποστήριξε την πρωτοβουλία αυτή. Το οριστικό σύστημα ΦΠΑ θα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις απώλειες ε, λόγω απάτης ΦΠΑ. Και φυσικά ε, δεν θα ε, διστάσουμε να υποστηρίξουμε τέτοιες προσπάθειες. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα για μας. Η Βουλγαρία δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ζημιών λόγω απάτης ΦΠΑ, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτή την ελευθερία ε, για να ε, πλουτίσουν παρανόμως μέσω του ΦΠΑ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν ε, να εξετάζουμε την τεχνική ανάλυση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την λεγόμενη ε, οδηγία εντάξει. Πριν βέβαια ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις ε, δεν μπορώ να σας μιλήσω για αποτελέσματα. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο στη διάρκεια της Προεδρίας μας. Όσον αφορά την διοικητική συνεργασία για θέματα ΦΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλέον παρουσιάσει την ανακοίνωσή της, τη συζητάμε και η Προεδρία θα κάνει προσπάθεια για να προχωρήσουμε και αυτό το ζήτημα. Εάν ε, τα καταφέρουμε, η διοικητική συνεργασία θα περάσει σε νέο επίπεδο. Θα υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ φορολογικών αρχών. Τον Οκτώβριο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της ε, και ε, υπογράμμισε κάποια σημεία για την εξυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος, για την καταπολέμηση της απάτης και την προσαρμογή του στην ψηφιακή εποχή. Εγώ πιστεύω ακράδατα στο σύστημα οριστικού ΦΠΑ ε, το οποίο θα μπορέσει να μας ε, ε, βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την απάτη Α και είμαι βέβαιος ότι και οι συνάδελφοι στο Συμβούλιο θα με υποστηρίξουν. you, Ο κύριος Φερνάντες, καλημέρα σας, καλώς ορίσατε ό,τι καλύτερο για την Προεδρία σας που μόλις αρχίζει και που σε οικονομικό επίπεδο έχει πολύ σημαντικές προκλήσεις μετά από τη δημοσίευση το Δεκέμβριο του Οδικού Χάρτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της Ευρωζώνης με αυτή τη μεταρρύθμιση του ESM, του European Stability Mechanism, και την εμβάθυνση. Ε, επομένως, σας περιμένει ένα συναρπαστικό εξάμεινο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, ε, ρωτήσω το εξής για την ολοκλήρωση του, ε, της Ευρωζώνης. Ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει την Τραπεζική Ένωση και προηγουμένως είχαμε εδώ τον ε, Εστονό Υπουργό ο οποίος μας εξήγησε πώς ε, προχώρησε η συζήτηση του κανονισμού που βρίσκεται ακόμα σε τεχνικό επίπεδο. Εσείς είπατε ότι αποτελεί προτεραιότητα για την Προεδρία σας και αυτό το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω είναι ποια είναι η στρατηγική της Προεδρίας σας ε, για να μπορέσουμε να αναβιώσουμε τις διαπραγματεύσεις ε, και πώς πιστεύετε θα μπορέσουμε να φτάσουμε και σε πολιτικό επίπεδο και ε, μέχρι να φτάσουμε στο πολιτικό επίπεδο, τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε να υπάρξει κάποια εξέλιξη στο τεχνικό επίπεδο και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε με την Τραπεζική Ένωση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γι' αυτό δεσμευόμαστε. Αλλά δεν αισιοδοξώ. Δεν ξέρω πότε θα λάβετε το ΙΔΙΣ. E Η συζήτηση στο Συμβούλιο είναι ακόμα στα σπάργανα. Σε τεχνικά πλαίσια φαίνονται όλα πολύ εύκολα. Μπορεί κάποιος να ε, συντάξει μια οδηγία. Υπάρχουν τρία επίπεδα προστασίας, τρεις πυλώνες, όλα αυτά είναι γνωστά. Αλλά ε, αυτό το οποίο δεν με κάνει να ευελπιστώ είναι το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη είναι αρκετά επιφυλεκτικά μεταξύ τους και νομίζω ότι εδώ πρόκειται για τη διαφορά βορρά-νότου. Οι χώρες του νότου θα ήθελαν να μειώσουν τους κινδύνους πρώτα και μετά να υπάρξει επιμερισμός κινδύνου. Υπάρχουν βέβαια και άλλες προσεγγίσεις, αλλά χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο χρόνο για συζητήσεις. Όπως σας είπα, θα συνεχίσουμε τις τεχνικές συζητήσεις. μαζί και με τον οδικό χάρτη του 2016, ε, βάσει και των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, αλλά να επαναλάβω ότι δεν αισιοδοξώ, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε πολιτικό επίπεδο σε ένα από τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν θα επανέλθει η σταθερότητα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και το θέμα αυτό. Μέχρι να γίνει αυτό δεν νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι. Σας ευχαριστώ. Περιμένουμε μια πιο επιθετική, για να τη χαρακτηρίσω έτσι, προσέγγιση για το φάκελο αυτό. Όλα αυτά βέβαια είναι θετικά και θα δούμε. Πρέπει και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Γιατί θα πρέπει και οι δύο εταίροι ε, να βρούνε κοινό τόπο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Βαντελάρε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε σήμερα και να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Έχω την εξή ερώτηση για το ΦΠΑ, γιατί ήθελα να πω το εξή Οι πρόσφατες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους διαφορετικούς συντελεστές. Εκεί συμφωνούν όλοι πως θα είναι πιο εύκολο να έχουμε έναν ενιαίο συντελεστή για κάποια προϊόντα και οι διαδικασίες ε, είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ αυστηρές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους συντελεστές ΦΠΑ παρουσίασε μια πρόταση όπου κάθε εθνική αρχή θα μπορεί να παρουσιάσει τις δικές της προτάσεις με τους δικές τους συντελεστές. Εσείς συμφωνείτε με την πρόταση αυτή ή θεωρείτε πως θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση έτσι ώστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αποφασίζεται σε ποια προϊόντα θα ισχύουν οι μειωμένοι συντελεστέ ΦΠΑ. Και επίση για το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα e-books θέλω να πω κάτι. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε και το 2017 και ξέρετε πως είναι ένα σημείο το οποίο είναι μπλοκαρισμένο στο Συμβούλιο γιατί δεν υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ της Τσεχίας και της Γαλλίας για το πώς θα γίνεται η αντίστροφη χρέωση. Αυτός ο μηχανισμός. Οπότε σας ρωτώ, εκεί τι γίνεται. Είναι δύσκολα τα θέματα αυτά και πώς να εξηγούμε εμείς συνέχεια στους πολίτες τι ισχύει. Οπότε στη δική σας Προεδρία Πιστεύετε πως αυτές τις δυσκολίες μπορείτε να τις ξεπεράσετε. Ξέρετε πως αυτή τη στιγμή άλλαξε η κυβέρνηση στην Δημοκρατία της Τσεχίας. Και επίσης, μία ακόμα ερώτηση. Ανησυχίες. Ανησυχίες πολλές έχουν εκφραστεί πως το ηλεκτρονικό βιβλίο και το ΦΠΑ, το ΦΠΑ στο σημείο αυτό θα συνδεθούν με το ευρύτερο, την ευρύτερη συμφωνία πακέτο για το ΦΠΑ. Εσείς πείτε μου, τα ηλεκτρονικά βιβλία θα τα βάλετε σε μια κατηγορία μόνο τους, εκτός αυτού του πακέτου που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, λοιπόν, ε, πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει κάποιες άτυπες επαφές και προσπαθούμε να κάνουμε μια διαμεσολάβηση μεταξύ Τσεχίας και Γαλλίας για το θέμα αυτό. Ναι, έχουμε νέα κυβέρνηση στην Τσεχία, αλλά ο υπουργό Οικονομικών, πρώην ε, υπουργό Οικονομικών είναι σήμερα Πρωθυπουργό και εκεί είχε ξεκινήσει όλη η συζήτηση με τη Γαλλία. Οπότε δεν βλέπω αν θα δείξει μεγαλύτερη ευελιξία. Το νέο πακέτο, να σας πω, για τον ΦΠΑ και το λέω αυτό μόνο ως εκπρόσωπος της Βουλγαρίας και Υπουργό Οικονομικών ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ στη Βουλγαρία και έχουμε μια έκθεση της Ernst Young με 250 σελίδες όγκο όπου αναφέρεται πως η μείωση συντελεστών ΦΠΑ σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων δεν, έχει καμία, δεν επηρεάζει καθόλου τις τιμές καταναλωτή. Εγώ δεν συμφωνώ με τους διαφορετικοποιημένους συντελεστές δεν νομίζω ότι αυτό είναι πλονέκτημα για τον τελικό καταναλωτή, μόνο διοικητικό βάρος προκαλεί, αλλά είναι εθνική απόφαση και αν η οδηγία επιτρέψει τέτοια ευελιξία στα κράτη-μέλη, είναι δικό του θέμα, εθνική πολιτική. Για μένα ο κατακαιρματισμός του ΦΠΑ και των συντελεστών αυτού δεν έχει καθόλου κοινωνική αξία, γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο πολύ εύκολα ξεπερνούν και χρησιμοποιούν συμπορικό πλεονέκτημα οι επιχειρήσει. Ναι, αλλά εθνική κυριαρχία και ευελιξία στα κράτη-μέλη είναι. Πάντα με βρίσκει σύμφωνο. Γιατί ο ΦΠΑ είναι ο βασικός, η βασική πηγή ο ίδιων πόρων για τα κράτη-μέλη και για του προπολογισμού, Οπότε αυτή η επιπλέον ελευθερία κινήσεων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να θεωρηθεί ω κάτι καλό. Και επαναλαμβάνω ω Βούλγαρο υπουργό Οικονομικών δεν σχεδιάζω να χρησιμοποιήσω αυτή τη δυνατότητα. Αυτή είναι η πολιτική μας. Και αυτό ισχύει εδώ και χρόνια. Το σύστημα ΦΠΑ στις Ευρωπαϊκές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλές φορές είναι απαρχιωμένο και τα κράτη-μέλη υποφέρουν από κακές αποφάσεις του παρελθόντος αλλά αν επιμένουν, εάν θέλουν να προσφέρουν αυτό το διαφοροποιημένο συντελεστή, κανένα πρόβλημα ο καθένας ό,τι πιστεύει. Πάντως, για τον τελικό καταναλωτή σας λέω πως δεν υπάρχει κανένα πλεονέκτημα. Αυτά είχα να πω. Thank you, Paul. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Ταν. Ευχαριστώ πολύ. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις περαιτέρω συζητήσεις και τη συνεργασία που θα έχουμε με την Βουλγαρική Προεδρία. τα δικά μου ερωτήματα σχετίζονται με ναι, τα αφορολογικά θέματα. Ε, όταν αναφερθήκατε στη διαφάνεια, ήρθε κατευθείαν στο μυαλό μου αυτό το ζήτημα των καταχώρα συστάσεων και των σχετικών εκθέσεων, ε, δηλαδή το κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί εδώ πρόοδο και κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ χρήσιμο, δηλαδή να επιτύχει η πρόοδος με αυτό το ζήτημα η Βουλγαρική Προεδρία. Επίση, αναφερθήκατε στην ενοποιημένη κοινή βάση εταιριών και ότι το ζήτημα είναι τεχνική φύση. Ε, ε, δεν νομίζω όμω, ε, κύριε Υπουργέ, πω έχετε δίκιο. Εμεί ε, ω Κοινοβούλιο δεν το εξετάσουμε ω ε, τεχνικό ζήτημα. Θα... Η συζήτηση θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο και θα είναι κατεξοχήν πολιτική. Οπότε θα ήθελα να μας πείτε πώς θα, ποια συνέχεια θα δώσει αυτή την τοποθέτηση που θα προκύψει από το κοινοβούλιο με αυτό το ζήτημα. Από εκεί και μετά. δύο ζητήματα. Νομίζω πως η Βουλγαρική Προεδρία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο και γνωρίζουμε πως η νέα κυβέρνηση συνασπού της Γερμανίας θα υποστηρίξει αυτή την, ε, αυτές τις προτάσεις. Οπότε ε, αν δεν υπάρχουν συστάσει του Συμβουλίου, καλό θα ήταν να υπάρξει μια τοποθέτηση από την πλευρά τη Βουλγαρική Προεδρία σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Είναι κέρια σημασία στο να προωθηθεί περαιτέρω αυτό το φάκελο και να φτάσουμε δηλαδή στην κατάλληλη, στην πιο σωστή αν θέλετε εναλλακτική. Και επίση ε, θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη αξιολόγηση των φορολογικών εισόδων των κρατών μελών. Ε, και προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό θα χρειαστεί συνεργασία από την Επιτροπή, μεταξύ της Επιτροπής αφενός και των ε, αρμόδιων φορολογικών αρχών αφετέρου. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκεντρώσει αυτά τα στοιχεία μόνη τη Επιτροπή. Οπότε θα ήθελα η Βουλγαρική Προεδρία να πιέσει, να ασκήσει πιέσει στα κράτη-μέλη έτσι ώστε πράγματι να ανταποκριθούν στη δική τους υποχρέωση ε, και να προβούν δηλαδή στις δικές τους εκτιμήσεις ως προς το τι θα σημάνει η κοινή ενοποιημένη ε, φορολογική βάση εταιριών ε, σε επίπεδο φορολογικών εσόδων. Υπουργό. Εγώ είμαι αισιόδοξο Ω προς το ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την κατάρθρον εξέταση του κειμένου διαβιβάζω το σχετικό κείμενο ε, στα κράτη-μέλη προκειμένου να ε, αποφασίσουν τελικά και να διαπιστώσουν κατά πόσο θα υπάρξει πραγματικά αντίκτυπο σε φορολογικό επίπεδο εφόσον πράγματι εφαρμοστεί αυτή η κοινή ενωπημένη φορολογική βάση εταιρεών. Σίγουρα η κοινή βάση θα είναι, θα είναι κέρια σημασία σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Ε, θα συμβάλλει δηλαδή θετικά σε αυτή. Στη Βουλγαρία έχει ξεκινήσει μια συζήτηση. Εμείς βέβαια έχουμε μια πολύ ευρία φορολογική βάση, δεν υπάρχουν δηλαδή κάποιες αντίθετες απόψεις, κάποιες αντιρρήσεις ε, σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Εμείς δηλαδή μόλις ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας σε ό,τι αφορά την φορολογική βάση Ε, θα προβούμε δηλαδή στην ενοποίηση όπως ε, προβλέπεται στο 3C ε, του κειμένου της οδηγίας. Τώρα σε ό,τι αφορά την πιο επιθετική εντός εισαγωγικών στάση μας απέναντι στα κράτη-μέλη ε, ακούω αυτό που μας είπατε σε ό,τι αφορά δηλαδή την αξιολόγηση στην οποία θα πρέπει να προβούν τις εφαρμογές αυτής της βάσης α, στα α, δημόσια οικονομικά τους. Ναι, ε, θα ήθελα επίση να σχολιάσετε το εξή, γιατί εγώ βρέθηκα μαζί με τον Αλένα Μασούρη στην δική σα χώρα και κάναμε κάποιε επικοδομητικέ συζητήσει. Ε, και ε, όσοι συναντήσαμε λοιπόν ήταν και πολύ καλά ενημερωμένοι αλλά εκείνο λοιπόν που θα ήθελα να μου πείτε είναι το, και που σα ρώτησα πολύ συγκεκριμένα ποια συνέχεια θα δώσετε στην τοποθέτηση του Κοινοβουλίου που το Φεβρουάριο Προφανώς θα λάβουμε υπόψη μας την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζουμε καλά ποιο είναι ο ρόλο που παίζει εδώ το Κοινοβούλιο. Και εγώ προσωπικά υποστηρίζω την CCCTB. Οπότε θα λάβουμε σοβαρά υπόψη την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου. Πρόεδρος, ε, ναι, προφανώς ε, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης θα ε, ληφθεί υπόψη και τοποθέτηση του Κοινοβουλίου. Κύριε Συνδεβά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ, με τα σχόλια που κάνατε και σε σχέση με το ΦΠΑ και σε σχέση με την κοινή βασική CCTB και να προσθέσω κάτι σε σχέση με τα όσα είπε μόλι τώρα ο Πολ. Λαμβάνοντα υπόψη δηλαδή τον ιδιαίτερα περίπλοκο χαρακτήρα τη διαδικασία του να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση σε ό,τι αφορά ε, την κοινή βασισή CCTB. Εάν δεν καταφέρουμε να φτάσουμε τελικά σε μια συμφωνία, μια ενισχυμένη συνεργασία, enhanced cooperation, θα μπορούσε να αποτελέσει μια βιώσιμη λύση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτή την ε, μετά στο κερδών ε, στο πλαίσιο δηλαδή της CCTB από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης, εγώ Είχα ε, συμμετάσχει σε εργασίε ε, ε, κεντρική ε, τράπεζα μα. Είχα δηλαδή, ήμουν επαγγελματικά ενεργό σε αυτό το τομέα και πραγματικά σέβομαι πολύ την προσπάθεια που κάνετε και την βούλησή σα να προσχωρήσετε στην ε, Ευρωζώνη. Αλλά ε, σε ό,τι αφορά την αύξηση του ΑΕΠ σα, Βλέπω πως ε, ο, τιμάριθμός σας, ε, ο πληθωρισμός δηλαδή, ε, αρχίζει να ανεβαίνει και δεν είμαι βέβαιος αν θα καταφέρετε τελικά να πληρώνετε το σχετικό κριτήριο για την προσχώρηση στην Ευρωζώνη, δηλαδή αυτή του, αυτό του χαμηλού ε, του πληθωρισμού. Σας ευχαριστώ. γνωρίζουμε πως η συνθήκη προβλέπει ορισμένες ε, δεσμεύσεις στο πλαίσιο δηλαδή της οθέτησης του ευρώ και βέβαια εδώ και 20 χρόνια βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία προσαρμογής μας ε, πράγματι ε, ο πληθωρισμός μας αυξάνεται λόγω ε, και των ε, παρόχων ενέργεια στη χώρα μας, αλλά είχαμε αντιμετωπίσει και προβλήματα αρνητικού ε, πληθωρισμού. Οπότε, τυπικά τη σημερινή ημέρα, εμεί πληρούμε το κριτήριο του πληθωρισμού. Και ακριβώς για αυτού τους λόγους υπάρχει και αυτή η διαδικασία της αναμονής, αν θέλετε, της πριν από την ένταξη στην Ευρωζώνη, τη μεταβατική, αν θέλετε, περίοδου. Άρα η δική μας ε, βούληση είναι να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, δηλαδή εκεί, αυτό το waiting room και να παραμείνουμε εκεί ε, μέχρι να είναι σίγουρο ότι πληρούμε όλα τα κριτήρια. Δεν θέλουμε δηλαδή να θεωρήσουμε, να προδικάσουμε ότι όλα τα κριτήρια πληρούνται. Τώρα, σε ό,τι αφορά την, ε, την της CTB. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία χαίρουν ορισμένων πλέον εκτιμάτων εντό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εγώ δεν θα χαρακτήριζα αυτή την κατάσταση ως ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών. Απλώς κάποια κράτη-μέλη είναι πιο επιφυλακτικά απέναντι ε, σε μια ταχεία εφαρμογή της ε, κοινή ενοποιημένης ε, φορολογικής βάσης των Παρ' όλα αυτά όμως, παρά δηλαδή αυτές τις ε, αμφιβολίες από την ε, πλευρά ορισμένων κρατών μελών, εγώ θεωρώ πως θα μπορέσουμε τελικά να κινηθούμε γρήγορα και πιστεύω πως ε, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε δηλαδή στο σχετικό κείμενο στο εγγύς Γνωρίζετε βέβαια πως θα πρέπει να υπάρξει ομοφωνία στο επίπεδο του Συμβουλίου και πράγματι υπάρχει ο κίνδυνος ένα και μόνο κράτος μέλος να μπλοκάρει την όλη διαδικασία. Ελπίζω όμως ότι θα καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο και σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Η ερώτησή μου αφορά την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ε, και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Οι προτάσεις είναι γνωστές, υπάρχουν οι προτάσεις του Κοινοβουλίου, υπάρχουν οι προτάσεις του Πρόεδρου της Επιτροπής του κ. Γιούγκερ, υπάρχουν και προτάσεις από τον Γάλλο Πρόεδρο τον κ. Μακρόν, η, προ... Ε, η Συμφωνία Προδιαπραγμάτευσης ε, για την ε, ε, κυβέρνηση του μεγάλου συνασπισμού στη Γερμανία. Ε, σταματώ τις παραθέσεις εδώ. Σε όλες τις περιπτώσεις αναφέρεται μια μεγάλη συμφωνία, μια συνολική συμφωνία που περιλαμβάνει μηχανισμούς μείωσης του κινδύνου και επιμερισμού του κινδύνου, μηχανισμού ευθύνη στον προπολογισμό και ε, δημοσιονομικής ευθύνης. Εσείς κάνατε κάποιες συγκεκριμένες αναφορές στην αρχική σας παρέμβαση και θα ήθελα απλώ να εμβαθύνετε λίγο περισσότερο ή δυνατόν. Πρώτον, Θεωρείτε εσείς αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ε, καλή συνεννόηση ως προς την το λεγόμενη μεγάλη συμφωνία ε, Ποιε είναι κατά την άποψή σα οι συγκεκριμένες πτυχές ε, τι οποίε θα πρέπει να ολοκληρώσουμε προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό ο οποίο θα έχει την απαραίτητη συνένεση ε, όλων των ευρωπαϊκών πρωτευουσών και φυσικά πώ βλέπετε το συγκεκριμένο ρόλο της ίδια σα της Προεδρίας για το θέμα αυτό. Να εξηγήσω καλύτερα τι εννοώ. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θεωρείτε ότι αποτελούν προτεραιότητα και μπορούν να υλοποιηθούν στη διάρκεια τη Βουλγαρική Προεδρία για να φτάσουμε πιο κοντά σε αυτή τη μεγάλη συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της νομισματικής ένωσης και την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης. Ευχαριστώ. θα προτείνουμε ένα προσαρμισμένο δικό χάρτη με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα βήματα για την ενίσχυση της Τραπεζικής Ένωσης. Προφανώς και χρειάζεται πολιτική συμφωνία, συνένεση σε πολιτικό επίπεδο. Ιδάλλως, οποιοδήποτε συμβιβασμός και οποιαδήποτε πρόοδος ε, δεν νομίζω να είναι δυνατός. Πιστεύω ότι στους επόμενους μήνες Μόλις έχουμε και κυβέρνηση στη Γερμανία. Θα υπάρχει περισσότερη επικοινωνία και διάλογος μεταξύ των μεγαλύτερων κρατών μελών και πραγματικά πιστεύω και ελπίζω ότι η Άντζελα Μέρκελ και ο πρόεδρος Μακρόν ε, θα προχωρήσουν το θέμα. Ως Βούλγαρος υπουργό ε, θα ήθελα να πω το εξής πριν υπάρξουν περαιτέρω δημοσιονομικές δυνατότητες για την Ευρωζώνη και πριν αποφασίσουμε κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει ένας Ευρωπαίος Υπουργός Οικονομικών, πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό και να αξιολογήσουμε πάρα πολύ καλά ε, τι θα μας προσφέρει αυτό και πού θα οδηγήσει, γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων όσον αφορά το, ε, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το ESM, ε, θα θέλαμε να επικεντρωθούμε στην ουσία της συζήτησης και όχι τόσο στην θεσμική σκοπιά για το Συμβούλιο, ανεξάρτητα από την προσωπική μου άποψη, αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει κάποια πρόοδος και να καταλήξουν σε μια κοινή θέση. Τα νομοθετικά κείμενα τα οποία θεωρούμε ότι μπορούμε ίσως ε, να προχωρήσουμε και να έχουμε κάποια πρόοδο είναι ο μηχανισμός σύγκλησης Πρόκειται για πάρα πολύ καλές πρωτοβουλίες ε, που ε, ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι αισιόδοξο λοιπόν. Μόλις υπάρξει κυβέρνηση στη Γερμανία νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ. Μπορούμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ καλή και επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με αυτή την νότα αισιοδοξία. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη. Πράγματι λοιπόν το εξάμεινο το δικό σας μπορεί να αποτελέσει κομβικό εξάμεινο ε, και να μπορέσουμε να κάνουμε τα αποφασιστικά βήματα για να προχωρήσει η νομοθεσία και το θεσμικό μας πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για τη δέσμευσή σας, συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία και ε, επικοδομητική συνεργασία στο εξάμεινό σας. Ευχαριστώ πολύ.